δεν ξέρω κατά πόσο όλοι πανηγυρίζουν τη συνθήκη της Λισαβόνας, τη θέση σε ισχύ. Ίσως πρέπει να μετακινηθούμε στο μπαρ και να βρούμε τους συναδέλφους να πίνουν σαμπάνια. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, διχασμένες απόψεις σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορώ όμως να σας πω ότι με τη θέση σε ισχύ η Ευρώπη θα μπει σε μια νέα εποχή όπου θα μπορούμε να ε, δράσουμε κατά πιο δημοκρατικό τρόπο και μεγαλύτερη διαφάνεια. Υπάρχουν ορισμένες προτινόμενες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν, και πρέπει να σας πω ότι κάπως με ενόχλησε αυτό, προτάθηκε να συζητηθεί ο αντίκτυπος της συνθήκης Λισαβόνας αύριο το πρωί αντί για σήμερα, διότι η Κομισιόν δεν έχει ε, ορίσει τα θέματα τα θέματα συναπόφασης που αφορούν τη συναπόφαση. Με εκπλήσει αυτό γιατί σήμερα το πρωί άκουσα στη... και διάβασα σε εφημερίδες ότι τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό και δεν κατανοώ γιατί δεν μπορεί να συζητηθεί την 1η ε, Δεκεμβρίου. Ελπίζω η συνεργασία μας να είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν, αρχίζοντας από αύριο. Άρα θα πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση για αύριο Ελπίζω όμως να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από την Κομισιόν που να μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Να λάβουμε τον κατάλογο λοιπόν από την Επιτροπή πριν από την έναρξη της συνεδρίας αύριο το πρωί. Μπορεί να μου το επιβεβαιώσει αυτό κάποιος. Φαίνεται πως όχι. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί, δεν μπορούμε να... γιατί πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση για αύριο τη στιγμή που δεν θα έχουμε ούτε αύριο τη λίστα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα είμαστε παρόντες αύριο. Ο Τζόναθαν, ο Τζόναθαν Φόλ θα παρευρίσκεται αύριο, αλλά δεν έχουμε τον κατάλογο έτοιμο σήμερα. Γίνονται συζητήσεις με την νομική υπηρεσία. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την νομική υπηρεσία. Ε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αλλά με εκπλήσει κάτι τέτοιο δεν κατανοώ γιατί δεν προετοιμαστήκατε νωρίτερα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνουν και οι εξής άλλες αλλαγές. Προτείνουμε να προσθέσουμε στη σημερινή μερίσια διάταξη την, ε, τη, τη συζήτηση των σημείων 13 με 18 για το πακέτο δέσμη μέτρων για το άσυλο και να αποσύρουμε την πρόταση ψηφίσματος ε, ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα. Επίσης ε, θα προσθέσουμε δύο σημεία. Η έκθεση Δίας Δεμέρα για την δημιουργία ενός δικτύου, ε, δικτύου σύνδεσης Σήμερα το πρωί θα συζητηθεί αυτό, καθώς και το SWIFT για αύριο το πρωί στις 10. Και εδώ νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος πολλών. Δυστυχώς το Συμβούλιο αποφάσισε για το SWIFT χτες, λίγες ώρες πριν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και υπάρχουν δύο χώρες που έχουν απόσχει και τη συγχαίρω γι' αυτό. Και θα ήθελα να προσθέσω τη δική μου πρόταση. Να έχουμε μία επεξήγηση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την κατάσταση όσο αφορά τις συμφωνίες PNR, προσωπικών δεδομένων δηλαδή των επιβατών με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία και φαίνεται ότι έχει επέλθει σύγχυση ως προς την, το, το νομικό καθεστώς που μας διέπει. Αυτό μας είπε η νομική υπηρεσία νωρίτερα. Θα πρέπει να ακυρωθεί η συμφωνία. Διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υφίσταται καν. Ζητήσατε το λόγο και τον έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ να εκφράσω και εγώ την ανησυχία μου και τη μεγάλη μου έκπληξη σε ό,τι αφορά και την καταγραφή της έκπληξης αυτής τα πρακτικά σε ό,τι αφορά τα θέματα της Λισαβόνας. Είναι δυνατό να μην τα συζητάμε τα πράγματα αυτά στην πρώτη συνεδρίαση, να μην είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τις αλλαγές αυτές στα πλαίσια της Λισαβόνας στην πρώτη συνεδρίαση. Χαίρομαι που το θέξατε το θέμα και θα πρότεινα η Προεδρία να ενημερώσει και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για την διαδικασία αυτή. Πώς αλλιώς να το δηλαδή, παρά περιφρόνηση, ως περιφρόνηση έναντι του Κοινοβουλίου, των Ευρωβουλευτών, του θεσμού του Ευρωκοινοβουλίου μετά από το παιχνίδι αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ασκήσω έντονη κριτική και να πω ότι χαίρομαι που το σχολιάσατε. Και το δεύτερο να πω ότι καλωσορίζω ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η Προεδρία έθεσε το θέμα του SWIFT στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα στο σημείο αυτό να προτείνω ο Πρόεδρος να φροντίσει κάποιος να παρευρεθεί από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου κατά τη συζήτηση που θα μας ε, παρουσιάσει και την νομική ε, κατάσταση από πλευράς του Κοινοβουλίου και κατά δεύτερον να παραβρεθεί και η Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να μας εξηγήσουν ποια είναι η θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Δεν θέλω να το συζητήσουμε τώρα επί του αύριο άλλωστε θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, απλά να τονίσω ότι αύριο θα πρέπει να συζητήσουμε με πάσα σαφήνεια πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία προκειμένου να υπάρχει καλή συνεργασία όντως. Ευχαριστούμε κύριε Στράσερ. Συμφωνώ πλήρως με τα σχόλιά σας και έχω καταγράψει τις υποδείξεις σας. Εξ ονόματος Προεδρίας αυτής της Επιτροπής θα κοινοποιήσω στον Πρόεδρο του Σώματος ότι η Επιτροπή δεν ήταν έτοιμη για την 1η Δεκεμβρίου. Και ε, θεωρώ ότι η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι παρούσα κατά τη συζήτηση του πακέτου SWIFT και θα ήθελα να προσθέσουμε αύριο το πρωί με την άδειά σας ότι θα ζητήσουμε μια διασάφηση για το PNR. Και εάν έχουμε κάποια διασάφηση εισήγηση μέχρι απόψε ή αργότερο το αργότερο αύριο το πρωί, θα ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο, διότι αν η συμφωνία PNR δεν ισχύει πλέον θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Γιατί τότε η μεταφορά δεδομένων είναι παράνομη. Συμφωνείτε με τις προσθήκες και αλλαγές που σας προανέφερα. Σχόλια όχι. Μιλώντας ε, για τη συνθήκη της Λισαβόνας, απόψε μετά την σημερινή συνεδρίαση στις 6.30 ο κύριος Λόπες, ο πρόεδρος της παρούσας επιτροπής, σας καλεί σε μια μικρή δεξίωση για ένα ποτό για τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και ελπίζω να πιούν μαζί μας και εκείνοι που δεν χαίρονται ιδιαίτερα ε, με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αλλά να πιούμε ένα ποτό όλοι. Συμφωνούντες και διαφωνούντες. Λοιπόν, έχω και κάτι άλλο να πω, αλλά νομίζω ότι αφορά τους συντονιστές. Θα ήθελα να δεχτείτε το διορισμό του κυρίου Κλάς από τους μη εγγεγραμμένους ως εισηγητή για τη συμμετοχή της ε, Ελβετίας και του Λίχτενστάιν στις δραστηριότητες του Frontex. Αντιρρήσεις όχι, ωραία, άρα αποφασίζεται. Τώρα προχωρούμε στο πακέτο στη δέσμη μέτρων για το άσυλο που προβλεπόταν για αύριο το πρωί, σημεία 13 έως 18. Και αρχίζουμε, συγγνώμη ένα λεπτό, διότι πρόκειται για πέντε εκθέσεις. Um, Φαντάζομαι ότι η χαρά και η ευθυμία μπερδεύουν ε, τον κατάλογο αγορητών. Καταρχάς έχουμε μία ενημέρωση για τα, τα ακόλουθα ζητήματα. κανονισμό του Δουβλίνου, οδηγία συνθήκων υποδοχής και ε, το Miss Eurodac. Αυτό θα μας το πει το Συμβούλιο από ό,τι μου είπανε. Ωραία. Δεν ξέρω ποιο, Ποιο θα μιλήσει από το Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μας δίνει την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τα νομοθετικά κείμενα που συζητώνται ή συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ειδικής παιδείας. Με πιάσατε κάπως εξαπίνης και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Νόμιζα ότι θα ξεκινούσαμε με την παρουσίαση των εισηγητών, αλλά τέλος πάντων ε, να ξεκινήσω, δεν έχω πρόβλημα να ξεκινήσω. Πώς έχει η κατάσταση. Χτε στο Συμβούλιο στην Υπουργική Σύνοδο είχαμε στην ημερήσια διάταξη μια ενημέρωση για την κατάσταση σε ό,τι αφορά την υποσυζήτηση νομοθεσία για θέματα ασύλου. Επίσης έγινε και μια παρουσίαση του, των νέων ε, προτάσεων για την οδηγία για τον καθορισμό του καθεστώτος πρόσφυγα και την οδηγία για τις διαδικασίες. Υποθέτω ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή θα συμπληρώσουν αυτά που θα πω σε σχέση με τις πρωτοβουλίες. Πρόκειται για νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής που δεν ε, συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Να μπω με τη σειρά που τα βλέπω στην ημερήσια διάταξή σας, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Συνθήκες υποδοχή. Uh, uh, Πρόκειται για μια οδηγία βέβαια που έχει στόχο να εξασφαλίσει το, υψηλό, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ε, αντιμετώπιση των ετούντων άσυλων σε ό,τι αφορά τι συνθήκε υποδοχή, την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων και την προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο των ε, δευτερογενών κινήσεων ε, των ετούντων άσυλων στα κράτη-μέλη. Έγιναν πολλές σχετικές συναντήσεις ήδη κατά τη διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας και η δική μας Προεδρία συνεχίζει το ίδιο έργο. Υπήρξε μεγάλη συμφωνία, ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποιες διατάξεις που παραμένουν συζήτηση. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κράτησης τώρα, της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και του ορισμού των μελών της οικογένειας. Σημειώνουμε επίσης ότι σε σχέση με τη γνωμοδότηση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο παραμένουν ακόμα κάποια ζητήματα όπου υπάρχει μία απόκληση των απόψεων και πάλι της πρόσβασης στην απασχόληση και το ζήτημα της κράτησης ε, εμφανίζεται όταν κάνει κανείς συγκρίσεις. Το Δουβλίνο. Η πρόταση αυτή δουλεύτηκε στις ομάδες εργασίας. Το βασικό εκρεμές ζήτημα και πάλι αφορά στον ορισμό των μελών της οικογένειας. Επίσης, είναι η διάταξη της προσωρινής αναστολής των μεταγωγών εν μέρει τα κριτήρια καθορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας οι διατάξεις για τις προσφυγές κατά των μεταγωγών και οι διατάξεις για την κράτηση καθώς και ορισμένες πτυχές του κεφαλαίου που ασχολείται με τις γενικές αρχές και τα εχέγγυα σε σχέση με άτομα που υποβάλλουν αίτημα διεθνούς προστασίας. Προχωρώντας τώρα στο Eurodac. Εδώ μπορώ να σας πω ότι υπήρξε αξιοσημείωτη πρόοδος. Uh, τα εκκρεμή ζητήματα σε επίπεδο Συμβουλίου αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένα το κύριο από αυτά αφορά στις διατάξεις πρόσβασης στα σχετικά, στις σχετικές πληροφορίες των διοπτικών αρχών. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση της περίοδου κράτησης αρχεία των δεδομένων των υπηκών τρίτων χωρών που ε, συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια τη διέλευση ε, των εξωτερικών συνόρων τη από δύο χρόνια σε ένα, η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών προτιμούν να κρατηθεί η διετή και όχι η ετήσια περίοδος. Αυτά για τις συνθήκες υποδοχής του Γιώργου και το Δουβλίνο. Θέλετε να συνεχίσω και με άλλες προτάσεις. Well, then I understand that uh, I could make uh, a short uh, Άρα να σας κάνω και μια σύντομη ενημέρωση για τις εργασίες της Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου και του κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να δώσω το λόγο στους συναδέλφους της Επιτροπής ως προς τα λοιπά. Το Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγράφουμε ότι υπήρξε βεβαίως ε, συμφωνία, υπάρχει και μια προγενέστερη κοινή θέση μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που είχε επίσης ε, συμφωνηθεί και το καταγράψει στην Επιτροπή σας. Πέραν αυτών, να σας ενημερώσω από τη χτεσινή συναντήση του Συμβουλίου ότι υπήρξε πολιτική συμφωνία ως προς την έδρα της, ε, του γραφείου αυτού. Συμφωνήθηκε μεταξύ των Υπουργών να πάει στη Βαλέτα. E uh, Σε ό,τι αφορά το κοινό πρόγραμμα εγκαταστασής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγιναν δύο συζητήσεις στο Συμβούλιο προχωρούμε προς την επιτεύξη συμφωνίας επί των βασικών αρχών για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Η Προεδρία είχαμε άτυπες επαφές με τους ορισθέντες εισηγητές της Επιτροπής σας και θα συνεχίσουμε βάσει των άτυπων αυτών συζητήσεων Προφανώς δεν υπάρχει ακόμα έκθεση από την Επιτροπή, ωστόσο επειδή επετέλεσε πολύ μεγάλη προτεραιότητα της Σουηδικής Προεδρίας να προχωρήσουμε στον τοσί αυτό, προσπαθούμε να εργαστούμε με τα κράτη-μέλη σε άτυπη βάση για να διευκολύνουμε την πορεία, την ταχεία πορεία της έκθεσης αυτής στην Επιτροπή για να ευθυγραμμιστούν οι απόψεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι στη φάση αυτή, αυτή είναι η πληροφόρηση του από πλευρά Συμβουλίου. Είμαι ανοιχτό σε ερωτήσει σα. Ένα εισηγητή ζήτησε το λόγο. Θέλετε να περιμένετε να μιλήσει η Επιτροπή. Όχι. Να, είπαμε να ρωτήσουμε πρώτα την Επιτροπή να μας κάνει μια παρουσίαση. Και μετά οι Κομισιόν ποιος θέλει το λόγο. να το καταλάβω. Δεν μπαίνουμε στι νέε προτάσει για, την υφιστάμενη, για τις θέλετε να μιλήσετε. Γιατί δεν σα άκουγα. Πώ Πώς έχει κατάσταση. Μα από ό,τι κατάλαβα θα μας κάνετε παρουσίαση και για τις νέες προτάσεις. Υπάρχουν πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεν τα κάνω όλα μαζί. Now, Καταρχάς, να συμπληρώσω αυτά που είπε η Προεδρία για το πώς έχουν τα πράγματα στις υφιστάμενες προτάσεις, στις υποσυζήτηση δηλαδή προτάσεις. Η Προεδρία υπογράμμισε ότι δεν είναι εύκολες στο Συμβούλιο Διαπραγματεύσεις στη συνθήκη, στην οδηγία της Συνθήκης υποδοχής. Η συζήτηση ήταν πραγματικά δύσκολες. Εγώ φαίνεται ότι είμαι κάπως λιγότερο αισιόδοξη από την Προεδρία. Πάντως υπάρχουν ε, σημαντικές αποκλήσεις μεταξύ της προτάσεως της Επιτροπής που είχε υποστηριχθεί ευρέως από το Κοινοβούλιο στην γνωμοδότησή του του Μαΐου. Το Κοινοβούλιο στην πράξη προσυπέγραψε όλες τις ε, αλλαγές που η Επιτροπή πρότεινε στην υφιστάμενη οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής και οι συζητήσεις στο Συμβούλιο, πώς να σας το πω, ήταν κάπως δύσκολες. Φαντάζομαι ότι, ο νέο, ότι η νέα επίτροπος θα εξετάσει το πώς θα προχωρήσει τον τομέα αυτό για να δει αν χρειαστεί να υποβάλει νέα τροποποιημένη πρόταση. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ωστόσο ακόμα. Περιμένουμε πρώτα να γίνει συζήτηση με τη νέα επίτροπο, γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Στην αγίωση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Για τον κανονισμό για το Δουβλίνο 2 υπάρχουν κάποια δύσκολα ζητήματα. Το είπε και ένα η Προεδρία. Οι συζητήσει ωστόσο συνεχίζονται. Η τελευταία ομάδα εργασία είπε ότι η Σουηδική Προεδρία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Υπάρχουν δυνατότητες συζητήσεων. Προχωρούμε αργά βέβαια. Για τον κανονισμό για το Eurodac, όπως ξέρετε, στην πρόταση αυτή υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η διάσταση τον άσυλο, αν θέλετε να την περιγράψω έτσι. Στο ζήτημα αυτό υπάρχει συνένεση του Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η άλλη διάσταση, η διάσταση των διοκτικών αρχών και εδώ πρέπει να λάβει θέση το Κοινοβούλιο, προφανώς. Και επίσης η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ε, έχει τεράστιες συνέπειες και αντίκτυπο σε, όλη, σε κάθε πρόταση τρίτου πυλώνα που κατά βάση είναι παροχημένη. Θα πρέπει η Επιτροπή να δει πώς θα προχωρήσει του τομεί αυτού. Ωστόσο τα θέματα είναι ακόμα υποσυζήτηση και δεν έχουμε οριστική θέση. Το ζήτημα αυτό επίσης θα πρέπει να συζητηθεί με την Επίτροπο όταν αναλάβει τις, τα καθήκοντα του χαρτοφυλακίου του επόμενο έτος. Αυτές είναι οι υποσυζήτηση προτάσεις. Να σας πω και δύο λόγια τώρα για, τη, για την οδηγία για τις διαδικασίες. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις. 21 Οκτωβρίου. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις διαδικασίες και της οδηγίας για τον ορισμό του πρόσφυγα. Ήταν τα δύο ελείποντα στοιχεία της δεύτερης φάσης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άρα η Επιτροπή υλοποίησε το καθήκον της να υποβάλει πρόταση αναμόρφωσης ολόκληρου του αρχιτεκτονικού συστήματος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου όπως το βλέπει και όπως είχε προγραμματιστεί στον προγραμματικό ε, στο, στο πρόγραμμα της Επιτροπής του 2008. Η οδηγία για τη συνθήκη για τις διαδικασίες. Ο κύριος στόχος της ε, πρότασης είναι να εξασφαλίσει υψηλότερα δυνατά επίπεδα προστασίας και μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης. Κάτι που θα έχει στόχο να μειώσει τις αποκλίσεις που υπάρχουν στο, στα ποσοστά αναγνώρισης ε, μεταξύ κρατών μελών εν ώψη τη δημιουργία μιας κοινή διαδικασίας ε, χορήγηση καθεστώτο πρόσφυγα όπω προέβλεπε το πρόγραμμα. Η πρόταση θέλει να διευκρινίσει, να απλοποιήσει, να ε, διαμορφώσει και να ενιώσει τις κοινέ ρυθμίσει για να βελτιώσει την ποιότητα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων ιδίω σε πρώτο βαθμό και να αυξήσει την ικανότητα των εθνικών αρχών να καταπολεμήσουν τις καταχρήσεις. Εν τέλει ήταν επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί συνέπεια με, την πρόσφατη, με τις πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας και στο ΔΕΚ και στο ΕΔΑ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πέντε ομάδες τροπολογιών που προτείνονται. Πρώτον, εν εισαγωγή ενιαίας διαδικασίας. Όλες οι αιτήσει κατά βάση διεθνούς προστασίονται υπό το φως και του ορισμού του πρόσφυγα και των λόγων επικουρικής προστασίας που παρέχει η οδηγία για τον ορισμό του πρόσφυγα. Δεύτερο πακέτο τροπολογιών. Εξασφάλιση καλύτερη, καλύτερης πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου. Οι προτινόμενες τροπολογίες θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητα των αρμοδίων αρχών να διακρίνουν μεταξύ ετούντων άσυλων και άλλων μεταναστών και να εφαρμόσουν τι συναφεί διαδικασίε γρήγορα. Αυτό πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό στα σύνορα τη Ένωση να αναγνωρίζονται πραγματικά και αμέσω αυτοί που έχουν ανάγκη διεθνού προστασία. Τρία νέα στοιχεία ε, προτείνονται σήμερα. Ένα. Οι αιτούντε άσυλο πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αιτήσει στι αρμόδιε αρχέ το συντομότερο δυνατό. Οι αρχέ δε έχουν ένα χρονικό περιθώριο 72 ώρων για να ολοκληρώσουν τις διατυπώσεις για την καταγραφή της αιτήσεως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, καθώς οι, οι υπάλληλοι των αρχών μετανάστευσης και φύλαξη των συνόρων συχνά είναι αυτοί που θα έρχονται σε, σε άμεση επαφή με τους ενδυνάμει ετούντες προστασία, θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά διαδικασιών που πρέπει πάντα να τηρούνται. Τρίτον, τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται επίση να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και τη συμβουλή για τι διαδικασίε ε, ασύλου στα σημεία εισόδου και στα σημεία κράτηση. Τρίτη ομάδα τροπολογιών, η ενίσχυση των κοινών δικονομικών εγγύσεων. Πρώτον, μείωση των υφιστάμενων εξαιρέσεων σε ό,τι αφορά τις βασικές εγγύησεις, ιδίω δε προτείνεται να εξασφαλιστούν ότι όλοι οι ετούντες έχουν τη δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης. Του, αυτή τη στιγμή σε κάποιες, υπό κάποιες περιπτώσεις ε, παρακάμπτεται η συνέντευξη. Επίσης θέλουμε να εισαγάγουμε επιπρόσθετες εγγυήσεις και ειδικέ δικλείδες ασφαλής για εξαιρετικά για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, θύματα βασανιστήριων ή θύματα σεξουαλικής βίας. Επίσης, να παρέχεται ε, δωρεάν νομική συνδρομή και βοήθεια στον πρώτο βαθμό. Οι τροπολογίες αυτές κατά την άποψή μας είναι ουσιώδεις για να εξασφαλιστεί το front loading πάνω στο οποίο ε, βασίζεται η πρόταση. Να βελτιωθεί δηλαδή η ποιότητα των πρωτοβάθμιων αποφάσεων, ούτω ώστε οι αποφάσει αυτέ να είναι αιτιολογημένες και αυτό θα βελτιώσει και την κατάσταση στα κράτη-μέλη, διότι θα υπάρχουν λιγότερε αποφάσει που ανατρέπονται στο δεύτερο βαθμό. Τέταρτον, επίσης εξετάζουμε το ενδεχόμενο μιας πιο ουσιαστική εφαρμογής του κεκτημένου ασύλου. Ε, ζητούμε να υπάρξει εξάμηνη διαδικασία για την ολο... περίοδος για την ε, ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας διαδικασίας. Αυτό, κατά την άποψή μας, επιτρέπει σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας να λάβουν τα δικαιώματα που τους χορηγεί η οδηγία για τον ορισμό του πρόσφυγα γρήγορα και όχι να περιμένουν για μεγάλο διάστημα. Ταυτόχρονα αυτό θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να απομακρύνουν γρήγορα όσους δεν χρειάζονται διεθνή προστασία. Επίσης, απλοποιούμε και ενοποιούμε τις διατάξεις για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης, προτείνουμε την διαγραφή της διάταξης που καθιστά δυνατή την υιοθέτηση κοινού καταλόγου χωρών, ασφαλών χωρών προέλευσης. Επίσης, επιτρέπουμε την ταχύτερη ε, διεκπαιρέωση των προδήλωσα βάσιμων αιτήσεων παραμένουν στη νέα πρόταση οι διατάξει αυτές για τους λόγους της αίτηση. Ε, πανεξετάζουμε ωστόσο την διάταξη για να δούμε μήπως μπορούμε να μειώσουμε την διαφοροποιημένη υλοποίηση από πλευρά κρατών μελών. Επίσης, εν τέλει ενισχύουμε τον όρο πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή. Οι τροπολογίες που προτείνουν προκύπτουν από την εξέλιξη της νομολογίας τόσο στο ΔΕΚ όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθετήθηκαν εν ώψη των διαδικασιών ασύλου. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι η αποτελεσματική προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου πρέπει να είναι και ε, για τα νομικά και για τα πραγματικά περιστατικά Εξετάζουμε τις εξελίξεις στι χώρες πρόέλευση και τρίτον και πιο σημαντικό, η πρόταση παρέχει ε, την γενική αρχή της αυτόματης ανασταλτικής ε, ε, εφαρμογής των προσφυγών. Θα σταματήσω εδώ. Αυτές είναι οι κύριες αλλαγές στην οδηγία για τις διαδικασίες. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο για την οδηγία για τον ορισμό του πρόσφυγα να είστε συνεπείς, αν γίνεται, για να μπορούν ε, να συζητήσουν το θέμα και τα μέλη. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Οι στόχοι της ε, πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για τον ορισμό του πρόσφυγα είναι εν γέννη παρόμοιες με αυτές που ανέφερε η συνάδελφος κ. Μαρτίνη. Κάποιοι βασικοί άξονες της αναθεώρησης αυτής. Πρώτον, διευκρίνηση κάποιων νομικών όρων για τον ορισμό των λόγων προστασίας βάσει μιας αξιολόγησης των λόγων που οδήγησαν σε κάποιες διαφορετικές αποκλήσεις ερμηνείας μεταξύ κρατών μελών. Πρώτον, ο φορέας προστασίας. Η πρόταση διευκρινίζει ότι η προστασία αυτή πρέπει να είναι αποτελεσματική και διαρκής και οι ε, προστασίας, οι μη κρατικοί φορείς προστασίας πρέπει να είναι και διατεθειμένοι να τηρήσουν το κράτος δικαίου και σε θέση να το κάνουν σε ό,τι αφορά την προστασία στο εσωτερικό της χώρας, την εσωτερική προστασία. Η πρότασή μας ήθελε να εξασφαλίσει κατά βάση την συμβατότητα της ε, διάταξης αυτής με την υλοποίηση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως έχει ερμηνευθεί σε μια πολύ πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑ η πρότασή μας ε, εισάγει τους βασικούς όρους για την εφαρμογή αυτή. Ο ετών πρέπει να έχει πρόσβαση στην συγκεκριμένη ζώνη και να λάβει την άδεια να εισέλθει και να εγκατασταθεί, καταργώντας τη δυνατότητα φυγής στο εσωτερικό της χώρας παρά τα, τα τεχνικά εμπόδια. Διότι αυτό θα ήταν ασύμβατο με τους ε, όρους που προανέφερα. Επιπλέον, η συμμετοχή σε μια κοινωνική ομάδα, ιδίως δε η διευκρίνηση ότι οι, οι διαστάσεις, οι έμφυλες διαστάσεις πρέπει να λαμβάνονται ε, υπόψη για να αποφασίσουμε κατά πόσον ένα άτομο μετέχει, αποτελεί ε, μέλος μιας κοινωνικής ομάδας υπό την έννοια της Σύμβασης της Γενέβης. Η πρόταση θέλει να βελτιώσει την αμφισημία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να εξασφαλίσει μια συνέπεια στην ερμηνεία των λόγων δίωξης, συνέπεια που προς το παρόν δεν διασφαλίζεται όπως το διαπιστώσαμε στην μελέτη αντικτύπου που συνοδεύει την πρότασή μας. Δεύτερο μεγάλο χαρακτηριστικό, η προσέγγιση των δύο καθεστώτων προστασίας. Η πρόταση καταργεί τους περιορισμούς των δικαιωμάτων των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Θεωρούμε ότι δεν είναι πλέον, δεν δικαιολογείται πλέον αντικειμενικά. Φερρυπίν, διάρκεια τίτλου διαμονής, πρόσβαση στην αγορά κοινωνική προστασία, η ε, υγειονομική προστασία, διατάξεις και ρυθμίσεις ένταξης. Τρίτον, διευκολύνουμε την ένταξη των δικαιούχων προστασίας. Αυτό ήταν ένα πολύ αδύναμο στοιχείο της εναρμόνισης της πρώτης γενεάς στον τομέα. Εμείς προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ένταξης που αφορούν ειδικά τους πρόσφυγες, διότι υπάρχουν πρακτικά εμπόδια στον τομέα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση ή σε μια σειρά διατάξεων και ρυθμίσεων ένταξης. Για παράδειγμα, επειδή δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία μια σειράς διπλωμάτων ή επαγγελματικής εμπειρίας. Πήγα γρήγορα, Πρόεδρε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να συνεργαστούμε με τους εισηγητές για τις δύο αυτές προτάσεις. Αυτό που συνάγω από τις προκατατικές συζητήσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης χτες είναι ότι υπάρχει μια γενική ικανοποίηση διότι με την κατάθεση των δύο αυτών προτάσεων η Επιτροπή θα επιτρέψει να γίνει μια πλήρης και περιστατωμένη συζήτηση για τα ζητήματα αυτά και ταυτόχρονα θα τηρούνται οι προθεσμίες που μας είχαν ε, τεθεί με βάση το σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου από τους ε, συνομοθέτες για την θέση σε εφαρμογή το 2012 το αργότερο των ε, ρυθμίσεων της δεύτερης γενεάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άννης Πλάσκαρτ έχει ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω οι άλλοι δύο εισηγητέ ε, είναι εδώ στην αίθουσα. Αν θέλει κανεί άλλο το λόγο, παρακαλώ να μα το ζητήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, σε ό,τι αφορά τι νέε προτάσει, τι καλωσορίζουμε, τι περιμέναμε και χαίρομαι που πλέον έχουν προταθεί και θα πρέπει να τα συζητήσουμε πολύ καλά αυτά στο Κοινοβούλιο και είναι σημαντικό να γνωρίσουμε και να δούμε ποιες είναι οι αρχές που προτείνονται στις προτάσεις. Έχουμε καθυστερήσει λίγο, όπως είπα και προηγουμένως, αλλά τι να γίνει τώρα επιτέλους μας υποβληθήκαν οι προτάσεις. Ευχαριστούμε το Συμβούλιο που έδωσε την έδρα στη Μάλτα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το βήμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο και αυτά που μας είπε, μου προκάλεσε έκπληξη αυτό που είπατε. Γιατί η συζήτηση για τους όρους υποδοχής έχει ήδη διεξαχθεί πολλές φορές. Και με ανησυχεί επίσης αυτό που είπε και η Επιτροπή για την Οδηγία για τους όρους ε, εισδοχής. Νομίζω ότι μια νέα τέτοια τροποποιητική πρόταση είναι απαράδεκτη, γιατί θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βγάλουν τελικά άκρη Άρα τι προτείνετε. αν ε, καταφέρει το Κοινοβούλιο να βρει μία λύση, το ίδιο θα πρέπει να κάνει και το Συμβούλιο για το Δουβλίνο. Θα συζητήθηκε καν χθε το Συμβούλιο. Μπορούμε να περιμένουμε όσο θέλετε, αλλά τελικά πότε θα σημειωθεί αυτή η πολύ αναμενόμενη πρόοδος. Σε αυτά θα περιοριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κανείς άλλος. Εξ ονόματος των δύο εισηγητών ίσων, ο κ. Μπουσουτήλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η κυρία Μάκοβεϊ δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί εδώ σήμερα το πρωί. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της. Δεν ε, υπάρχουν μεγάλα εκρεμή αμφιλεγόμενα ζητήματα τα οποία να, χρειάζω, να χρειάζεται να τονίσουν να υπογραμμίσω εξ ονόματος της. Να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις Κοίταξα και εργάστηκα επί της πρότασης χτες σε ό,τι αφορά το γραφείο ασύλου. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν επηρέασα καθόλου την απόφαση, αλλά χαίρομαι που το γραφείο θα ιδρυθεί πλέον στη χώρα μου. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που πλήττουν ε, τις νότιες χώρες, αλλά νομίζω ότι αποτελεί και ένα μήνυμα για τα ίδια τα κρατη για να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά θα στρωθούν στη δουλειά και θα κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Στον ίδιο βαθμό λοιπόν που θέλω η Ευρώπη να βοηθάει χώρες όπως η δική μου, θα ήθελα και τα μέλη, αν θέλετε, τις νότιες χώρες να κάνουν και αυτές το μερίδιό τους της δουλειάς. Σε ό,τι αφορά την ατζέντα τώρα για το Γραφείο Ασύλου επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον, την, Jean, ε, την, την, την Jean Lambert. Δεν ξέρω αν είναι εδώ σήμερα, αλλά πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά για να πετύχουμε το συμβιβασμό με το Συμβούλιο και προφανώς και τις αξίζουν έπαινοι για τα διάφορα στοιχεία τώρα στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να πω ότι λυπάμαι που φαίνεται ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόοδος στο εσωτερικό του Συμβουλίου για τα διάφορα στοιχεία και όντως γιατί αφαιρέθηκε το γραφείο ασύλου από το όλο πακέτο ασύλου γιατί ήταν η πιο απλή πρόταση επί της οποίας μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στο ιστορικό του Συμβουλίου και φαίνεται ότι όλες οι άλλες προτάσεις ε, αποτελούσαν δύσκολα θέματα για το Συμβούλιο. Και όπως και η Ζανίν, θα ήθελα το Συμβούλιο να κατέβαλε μεγάλη, μεγαλύτερη ε, προσπάθεια σε ό,τι αφορά τις ε, δυσκολίες επί της ουσίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Δουβλίνου όπου σαφέστατα εκεί κολλάει το όλο σύστημα και θα πρέπει να καταπιαστούμε με τα θέματα αυτά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Για τη νέα πρόταση τώρα, για τις νέες προτάσεις μάλλον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της και νομίζω ότι ως Επιτροπή, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να επισέλθουμε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας, αν θέλετε, να εξετάσουμε πολύ λεπτομερώς, πολύ εντελεχώς τις προτάσεις αυτές. Πρόκειται για προτάσεις κλειδιά για την ε, διαμόρφωση μιας κοινή ε, πολιτικής για το άσυλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να τις εξετάσουμε εντελεχέστατα. Θα πρέπει προφανώς σε πρώτη φάση ως Επιτροπή να ορίσουμε εισηγητή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και όταν θα έχει γίνει αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τις προτάσεις ε, λεπτομερώς για να βεβαιωθούμε ότι θα είναι συνεκτική και σωστή η άποψη που θα παρουσιάσει στην πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Μπουσουτή, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτές τις τελευταίες προτάσεις θα πρέπει να λεφθούν υπόψη και να εξεταστούν από τους συντονιστές σε ό,τι αφορά τον ορισμό του εισηγητή και την διοργάνωση ίσως ακροάσεων. Για να το βάλουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ, Σοφή. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι ο Αντώνιο Χιντάλικο δεν μπορεί να παρευρεθεί ο εισηγητή, γιατί άλλαξε η μερίσια διάταξη. Αυτό προκαλεί μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι θέλει να θέσει κάποια σε μια κλειδιά αύριο στη συζήτηση. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τη Ζανίν. Πλέον το πακέτο έχει τεθεί σε κίνηση. Είναι προφανές ωστόσο ότι για το θέμα των διαδικασιών, των γυροντάκτη ε, του Δουβλίνου, όλα αυτά τα δύσκολα θέματα δεν έχουν σημειώσει η πρόεδρο. Να σας πω για τη Eurodac για παράδειγμα, ότι το Συμβούλιο ανέφερε το θέμα της πρόσβασης σε βάση δεδομένων από τις αρχές εφαρμογής του νόμου. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα, τα αμφιλεγόμενα και από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μα είπατε δεν έχει σημειωθεί καμία απολύτω πρόοδο στο σημείο αυτό. Και έχει δίκιο ο Σάιμον. Θα πρέπει να συγχαρούμε την Τζιν Λάμπερτ και το Γραφείο Ασύλου. Αφαιρέθηκε το θέμα αυτό από το πακέτο γιατί ήταν το εύκολο αν θέλετε σημείο και ευτυχώ καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ότι πλέον θα εντρεθεί αλλά έχουμε πολύ πιο δύσκολε διαδικασίε με το Δουβλίνο πλέον με του όρου ε, εισδοχή. θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά για να περάσουν για τα πακέτα αυτά. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω και την εορταστική ατμόσφαιρα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αλλάζουμε την ατζέντα. Αυτό δεν ε, συμβάλλει, αν θέλετε, στην όλη πρόοδο του θέματος. Και τέλος να συγχαρώ την Μάλτα και τον Σάιμον και επίσης αν δεν λειτουργεί στο γραφείο, ξέρουμε ποιον θα κατηγορούμε πλέον. Ο Σάιμον, μεγάλη η ευθύνη που σε βαραίνει πλέον. Μάλιστα. Πρωτού δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Ταβάρη. Συμφωνώ με τα σχόλιά σα για την αλλαγή της ημερησία διάταξη. Χτες με ενημέρωσαν το βράδυ, μην νομίζετε. Ε, με ενημέρωσαν, δεν με ρώτησαν και με ενόχλησε ιδιαιτέρως και με ενόχλησε ακόμα πιο πολύ το γεγονός ότι σήμερα το πρωί ανακάλυψε ότι η αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είχε καταφέρει να προετοιμαστεί για τη συνεδρία σε τη σημερινή και υπέθεσα εσφαλμένα ότι είχαν ενημερωθεί και οι συγητές για τις αλλαγές αυτές την ημερήσια διάταξη και με μου προκαλεί ιδιαίτερη ενόχληση το γεγονός ότι προφανώς δεν ειδοποιήθηκαν και τι να σας πω, φαντάζομαι ότι όλοι μας ενοχλούμαστε. Γιατί όλοι μας έχουμε γεμάτες ημέρες, προσπαθούμε να τις οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μας συμφωνείτε μαζί μου ότι τέτοιες αλλαγές δεν θα πρέπει να γίνονται παρά μόνο αν έχουμε όλοι ενημερωθεί εγκαίρως και αν υπάρχει σοβαρός λόγος, αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Γιατί φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενημερωθεί και πριν από χθες το βράδυ σχετικά με τους λόγους που προκάλεσαν την καθυστέρηση αυτή. Ο κύριος Ταβάρης. Well, uh, Φαίνεται ότι όλοι μιλούν, μιλούν αγγλικά. Σήμερα δεν θα το κάνω, διότι σήμερα είναι η Ιερά Μέρα στην Πορτογαλία, διότι έχουμε την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας μας. Ε, άρα δεν μπορώ παρά να μιλήσω πορτογαλικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι οι δέσμοι μέτρων για το άσυλο και θα ήθελα να πω ορισμένα λόγια επί του θέματος, αλλά δεν είναι το θέμα προς συζήτηση. Ωραία. Περνώντας στα πορτογαλικά θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την απόφαση που ελήφθη σε σχέση με το γραφείο τη... στη Μάλτα. Η συνάδελφος Jean Λάμπερτ εργάστηκε πολύ σκληρά για αυτό το πακέτο, έτσι ώστε να υπάρξει μια παγιοποίηση της κατάστασης και νομίζω ότι αυτό αποτελεί καλό δείγμα για τις συζητήσεις που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μετανάστευση και για τη χορήγηση ασύλου, διότι υπάρχουν μεγάλες διχογνωμίες και σε επίπεδο κοινή γνώμης ε, σε σχέση με το ποια στάση θα πρέπει να λάβουμε ως προς τα μεταναστευτικά φαινόμενα και τις μεταναστευτικές ροές και πέρα από αυτές τις μεγάλες διαφορές ε, δεν έχουμε ανταγωνιστικές θέσεις. Δεν εμένουμε σε ανταγωνιστικές θέσεις και προσπαθούμε να προωθήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική έναντι του φαινομένου της μετανάστευσης. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να φτάσουμε σε νέες συνενέσεις μεταξύ χωρών του Νότου και, της, και του Βορρά, καθώς και της δεξιάς και της αριστεράς στο σώμα αυτό. Είναι πολύ καλό το νέο αυτό, το οποίο δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά και πιστεύω ότι το άσυλο και η μετανάστευση δεν πρέπει να αφορούν μόνο τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών και πρέπει να δημιουργηθούν και άλλοι φορείς σε επίπεδο Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Αρρωγής και Μετανάστευσης, εκεί που υπάρχουν οι Υπουργεία Μετανάστευσης, έτσι ώστε να μην μιλάμε μόνο για συνεργασία, για διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σε σχέση με την δέσμη μέτρων για τη χορήγηση ασύλου. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα ενδιαφέρον φαινόμενο και προσπάθεια εναρμόνισης των διαφόρων φορέων που σχετίζονται με τη χορήγηση ασύλου έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Αλλά το πακέτο δεν είναι εξισορροπημένο. Έχουμε μεγάλο βαθμό λεπτομερίας σε ορισμένες τυχές, αλλά υπάρχουν και ορισμοί οι οποίοι είναι αρκετά συγκεχημένοι και οδηγούν σε αυθαίρετα συμπεράσματα, τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν δημοκρατικά και να επαληθευθούν δημοκρατικά. Γι' αυτό νομίζω ότι οι συγητές θα πρέπει να καλύψουν αυτά τα κενά. Το ένα παράδειγμα που θα σας δώσω σχετίζεται με την πληροφόρηση. Δεν υπάρχει στην ουσία πληροφόρηση σε σχέση με τους ετούντες άσυλο. Δεν ξέρουν δηλαδή τι δικαιώματα έχουν και νομίζω ότι θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και σε σχέση με τις ιατρικές εξετάσεις κατά την ε, ε, εισδοχή σε ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχουν ορισμένα βασικά κενά και είναι γεγονός ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διενεργήσουν ιατρικές εξετάσεις, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά ότι δεν χορηγούν άσυλο, ακριβώς επειδή οι αιτούντες άσυλο δεν υποβλήθησαν σε ιατρικές εξετάσεις. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά είναι γεγονός ότι το γραφείο αυτό αποτελεί μια πολύ καλή ε, δημιουργία και πιστεύω ότι όπως είπε η Τζιν Lambert, θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος των φορέων και των θεσμικών οργάνων και η πραγματικότητα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας επιβάλλει από το Κοινοβούλιο να ηγείται αυτή τη διαδικασία σε σχέση με το δημοκρατικό μα έλλειμμα και τον δημοκρατικό έλεγχο ο οποίο επιβάλλεται. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Στράσερ και μετά η κυρία Φλότρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να σας συγχαρώ για την πρόταση για το γραφείο υποστήριξης και για την απόφαση που ελήφθησε. Είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό προς την κατεύθυνση εναρμόνισης και είναι σημαντικό το ότι τελικά θα τρέψει στη Μάλτα, ένα από τα βασικά προβληματικά σημεία της Ευρώπης και ελπίζουμε λοιπόν ότι πολύ γρήγορα θα αναλάβει τη δράση του και τη λειτουργία του το γραφείο αυτό. Νομίζω ότι στο παρόν, ε, στην παρούσα φάση της συζήτησης το θέμα δεν είναι να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αλλά τις βασικές γραμμές που συνδέουν όλες αυτές τις οδηγίες ή θα έπρεπε να τις συνδέουν. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω δύο βασικές γραμμές ε, επιτάπητος που με απασχολούν ιδιαίτερα. Καταρχάς θα ήθελα να καλέσουμε και εμπειρογνώμονε οι οποίες θα α, ελέγξουν τα προτινόμενα μέτρα. Γιατί αυτοί τελικά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αυτοί θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα προκύψουν αν δεν λειτουργήσουν σωστά τα μέτρα μας. Και έχω την αίσθηση ότι ίσως κάποια πράγματα τα οποία προτείνονται με καλή πρόθεση για να απλοποιήσουν την κατάσταση, τελικά συνεπάγονται τεράστιο κόστος και τεράστιο γραφειοκρατικό άχθος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε. Κατά δεύτερον, η εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών προκειμένου να προκύψει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Εντάξει, όχι όμως να γίνει κεντρική διαμόρφωση Νομίζω ότι δεν συμφέρει κανένα να προδιαγράψουμε λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στη Μάλτα, όπως και στην Πολωνία, στη Σλοβακία. Όχι, χρειαζόμαστε γενικές κατευθυντήριες γραμμές, χρειαζόμαστε ανώτατα και κατώτατα όρια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε ξεχωριστή κατάσταση το κάθε κράτος μέλος να έχει ένα περιθώριο δράσης. Γιατί αν προσπαθήσουμε όλα να τα ρυθμίσουμε από τις Βρυξέλλες, πραγματικά δεν θα έχουμε επιτυχία. Ευχαριστούμε κύριε Στράσερ, η κυρία Φλότχ και μετά η κυρία Λάτσφορντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είχα ήδη την ευκαιρία να πω ότι το πακέτο ασύλου πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση ένα, αλλά πολύ μακριά ήμασταν ακόμα για να υπάρξει μια πλήρης ευρωπαϊκή ή διεθνής προστασία στο ύψος των δεσμεύσεων και των φιλοδοξιών μας. Διότι η συνέπεια με τέτοια διεθνούς προστασίας απαιτεί κατά την άποψή μου την κατάργηση των συμφωνιών του Δουβλίνου που έχει πραγματικά επαχθέστατες συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του ασύλου στην Ευρώπη, ιδίω διότι πολλοί Πολλά άτομα που δεν βρίσκονται πλέον στην πρώτη χώρα άφηξή του στην Ευρώπη αρνούνται να ζητήσουν το άσυλο εκεί, φοβούμενοι να επιστρέψουν στη χώρα αυτή. Άρα το άσυλο, ένα άσυλο άξιο του ονόματό του στην Ευρώπη, η ικανότητα, περιλαμβάνει και την ικανότητα του ατόμου να επιλέξει τη χώρα ασύλου στην οποία θα μπορεί να ενταχθεί με περισσότερη επιτυχία για λόγου ιστορικού, οικογενειακού, φιλικού κλπ. Επίση, η αμοιβαία αναγνώριση Τη ικανότητα ε, να κυκλοφορήσουν ελεύθερα τα άτομα που αναγνωρίζονται σε μια χώρα τη Ευρώπη και αλλού. Το πακέτο πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση όπω σα είπα, αλλά βρισκόμαστε μακρά της πλήρου επιτυχίας. Μια συγκεκριμένη ερώτηση προ την Κομισιόν. Καταλαβαίνω και εγκρίνω την ιδέα να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την ε, επαναπρόθεση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Άρα χρειάζεται να υπάρχει ενημέρωση όλων για την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Αν είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να, να βρούμε μεταξύ των πιθανών μεταναστών όσους χρειάζονται διεθνή προστασία. Και τους άλλους, όπως σωστά είπατε, να μπορούμε να τους επαναπροωθήσουμε γρήγορα. Εγώ σας ρωτώ, τι προβλέπετε συγκεκριμένα για να καταστεί αποτελεσματική μια τέτοια απόφαση. Διότι η κοινή εμπειρία μας, όσοι ξέρουν τις διαδικασίες αιτήσεων ασύλου στι πατρίδε τους, είναι ότι αν δεν υπάρχουν ανεξάρτητα όργανα, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που είναι δραστηριε στον τομέα, αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι επαρκώ καταρτισμένοι και με σεβασμό των ε, δικαιωμάτων των μεταναστών και των ετούντων άσυλων, πολύ λίγες πιθανότητες υπάρχουν να υπάρξουν ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τι προβλέπει λοιπόν η Κομισιόν για να καλύψει το ζήτημα αυτό. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τις δραστηριότητες Frontex στη θάλασσα. Τι γίνεται για να σταματήσει να υπάρχει συστηματική ε, αποτροπή σκαφών προ τη Λιβύη ή την Τουρκία. Κάτι αρκετά κοινό και μάλιστα με άγριο τρόπο από πλευρά ορισμένων χωρών. Η Σάρα Λάτφορντ. Ευχαριστώ. Κάποιες σκέψεις για το Eurodac. Από σήμερα δεν θα έχουμε πλέον μέτρα πρώτου και τρίτου πυλώνα. Και άρα δεν θα υπάρχει διαχωριστική αντιμετώπιση των μέτρων ασύλου του πρώτου πυλώνα και της διοκτικής προσέγγισης του τρίτου πυλώνα. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την όλη διαδικασία του, του Eurodax. Στην πραγματικότητα, Όταν χρειάζεται μια μεθοδιακή δράση, χρειάζεται εμπλοκή της διοκτικής αρχής. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να εξετάζουμε από την αρχή ζητήματα αναλογικότητας και να λαμβάνουμε υπόψη το ότι η το και στο εξή αστυνομία θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του γιοντακ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, από την οπτική γωνία του πρώτου πυλώνα κάναμε καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και μετά να το ανατρέπουμε αυτό από την οπτική γωνία του τρίτου πυλώνα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ας μην ε, βαφκαλιζόμαστε. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Και μετά από την απόφαση του δικαστηρίου για το DNA πριν από ένα χρόνο και της ανάγκης να λειτουργούμε με βάση την αρχή της αναλογικότητας σε μια δημοκρατική την ε, αναλογικότητα της ε, νομοθεσίας. Μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία αυτά, όπως και άλλα τα PNR, ας πούμε το SWIFT, δεν συλλέγονται κατά βάση και καταρχήν για τη χρήση από τις διοκτικέ αρχές, αλλά για άλλους λόγους. Λοιπόν, να το ξαναδούμε από την αρχή. Θέλει κανένας άλλος το λόγο για να κλείσουμε. Κύριε Ματιέ. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη για την τοποθέτηση του γραφείου στη Μάλτα. Μπορεί να μην ε, είναι αρμόδιος, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το συγχαρούμε ούτως ή άλλως τον κύριο Μπουσουτήλ. Μία διευκρίνηση θέλω από την Επιτροπή για το άσυλο. Θα περίμενε εναρμόνιση. Αυτό είναι θετικό. Και θα ήθελα μια διευκρίνηση για την έννοια της, ε, των μελών της οικογένειας. Κομισιόν, μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που τέθηκαν. Δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τα χρονικά μας όρια, αλλά πραγματικά είμαστε στο τσάκ. Λοιπόν, να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, Δεσποινής. Προεδρίνα. we will um, use new words very briefly on the last question για το τελευταίο αυτό ερώτημα να σας απαντήσω για τον ορισμό της οικογένειας δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείται δεν κατάλαβα τι ακριβώς ε, εννοείται τι συμβαίνει στα μέλη της οικογένειας, δηλαδή ποια είναι ο ορισμός, ποιες είναι οι προτάσεις ή οι τροποποιήσεις που προτείνονται, αυτό εννοείται. Εγώ έτσι καταλαβαίνω την ερώτηση, κυρία Ματιό. Θα θέλατε να διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείται. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ορίζεται την επανένωση της οικογένειας. Πώς ορίζεται η οικογένεια. η Επιτροπή πρότεινε κάποια τροποποίησεις στον ορισμό της οικογένειας από το πρώτο είδη πακέτο το οποίο παρουσιάστηκε πέρσι και επιλέξαμε μία συνεκτική προσέγγιση για όλη την πρόταση. Δεν άλλαξε δραματικά ο ορισμός της οικογένειας, είναι δύσκολο το θέμα αυτό όπως γνωρίζετε. Ωστόσο, προτείναμε προτείναμε να ληφθούν υπόψη μέλη της οικογένειας ανήλικα αλλά που έχουν παντρευτεί όταν είναι προς το συμφέρον τους. Εξαρτάται από τους όρους της οικογένειας και επίσης προτείναμε να συμπεριληφθούν τα ανήλικα αδέρφια παντρεμένα ή μη εφόσον είναι προς το συμφέρον τους. Αυτές ήταν οι βασικές αλλαγές που προτείναμε στον ορισμό της οικογένειας οι οποίες ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την αποδοχή από το Συμβούλιο, από τα κρατη ιδιαίτερα στο πρώτο πακέτο, άρα δεν περιμένω καλύτερη τύχη για το δεύτερο, τη δεύτερη πρόταση για το θέμα του Δουβλίνου τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πέρα από τον ορισμό της οικογένειας που έχει λίγο διευρυνθεί για να μην υπάρχουν καταχρήσεις, για να είμαστε ρεαλιστές, προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε κάποια από τα κριτήρια για την επανένωση με μέλη της οικογένειας και με συγγενείς, προκειμένου να διευκολύνεται η επανένωση οικογένειας στο Δουβλίνο. Αυτό είναι ένα θέμα για τα θέματα τα οποία έθιξε η κυρία Φλότρ. Δεν θέλω να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, ωστόσο στην παρουσίασή μου προσπάθησα να επισημάνω κάποιες από τις αλλαγές οι οποίες κινούνται όλες προς την κατεύθυνση που υποδείξατε σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των συνόρων, την εφαρμογή της κατάρτισης, της πρόσβασης της διαδικασίας. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία Μάλλον ένα στοιχείο το οποίο θέλαμε να τονίσουμε είναι η πρόσβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικτές ροές, που είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Η νομική αρρωγή σε πρώτη... Σε πρώτη φάση λοιπόν, μιλάμε για δωρεάν νομική αρρωγή εξ αρχής, όχι όταν έχει ληφθεί η απόφαση. Πρόκειται για μια καινοτομία που δεν υπάρχει δεν προβλέπεται από κανένα μέσο γιατί υπάρχει νομική αρρωγή όταν έχει ήδη ληφθεί μία απόφαση κατά ενός ατόμου και θέλει να ασκήσει έφεση το άτομο αυτό. Όχι, τώρα μιλάμε για νομική αρρωγή εξ αρχή. Και αναφέρω μόνο δύο σημεία, θα μπορούσα να συνεχίσω. Και όπως είπε και ο κύριος Μπουζουλτήλ, μιλάμε για πολύ περίπλοκα εργαλεία. Χρειάζεται λοιπόν πολύ πιο λεπτομερή συζήτηση και χρειάζονται πολύ πιο λεπτομερείς ε, ερωταπαντήσεις. Ιδάλλως μπορώ να συνεχίσω επαόριστο να μιλάω για το θέμα του Frontex τώρα. Είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Νομίζω ότι τα περιστατικά δεν που αναφέρεται δεν αποτελούσαν επιχειρήσεις Frontex, αλλά κάποιον κρατών μελών. Δεν νομίζω ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του Frontex, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί μου ζητήσατε να είμαι και σύντομη. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Το Συμβούλιο θέλει να προσθέσει κάτι ή θεωρείτε ότι σας καλύψαν. Εντάχει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας σε σχέση με την απόφαση της έδρας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό και θα ήθελα να σας πω ότι ο Υπουργός μου ε, θα παρευρεθεί εδώ στις 7 του μηνός για να συζητηθούν τα αποτελέσματα της Σουηδικής Προεδρίας σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να σταθεί σε αυτό, διότι ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα της Σουηδικής Προεδρίας. Ως προς το θέμα της περιορισμένης προόδου στα, στη δέσμη μέτρων για το άσυλο, εμείς ως Σουηδική Προεδρία ήμασταν θύματα του γεγονότος ότι υπάρχουν πολλά, πολύ αλληλένδετοι φάκελοι και ήταν δύσκολο ε, να προωθήσουμε ορισμένους φακέλους τη στιγμή που οι αντιπροσωπείες ξέρουν ότι οι φάκελοι αυτοί θα υπάρχουν σε περχόμενες προτάσεις. Γι' αυτό είχαμε περιορισμένη πρόοδο. Έχει επιτελεστεί πρόοδο σε μεμονωμένα θέματα και αφορούν τις προτάσεις που βρίσκονται επιτάπητος και εδώ έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν πραγματικές διχογνωμίες στο Συμβούλιο μεταξύ κρατών μελών και ορισμένα, ορισμένοι βουλευτές αναφέρθηκαν στο γεγονός αυτό. Αυτό το παρατηρήσαμε αρκετές φορές στο Συμβούλιο και σε πολιτικό και υπουργικό επίπεδο ε, έχουν εκδηλωθεί. Ως προς τα σχόλια του κυρίου Στράσερ θεωρώ ότι με την καθιέρωση ενός γραφείου υποστήριξης. Θα το δούμε από πρακτική πλευρά περισσότερο, από πλευρά εφαρμογής δηλαδή, διότι τότε οι κυβερνήσεις, η δημόσια διοίκηση των κρατών μελών θα δούμε τι θα κάνει σε καθημερινή βάση. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και αυτό το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης και αυτά ήταν τα σχόλια μου. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Άρα τελειώνουμε με αυτή τη συζήτηση ως προς τη δέσμη μέτρων για το άσυλο. Ορισμένα μέλη μίλησαν, μάλλον εκφράστηκαν αρνητικά για την έλλειψη προόδου και δεν πρόκειται για ορισμένους μόνο βουλευτές. Απλώς όλοι θα περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη ε, προόδο όχι τους δύο τελευταίες, τελευταίους μήνες, αλλά στην τελευταία δεκαετία. Θα ήθελα λοιπόν το Συμβούλιο να προωθήσει το ζήτημα ενεργά, ακόμα και αν έχει λάβει μία σωστή απόφαση καταρχήν. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μακρύς ο τίτλος. περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλκάιδα και του Ταλιμπάν σε σχέση με τη Ζιμπάμπουε και κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών εν ώψη της κατάστασης στη Σομαλία. Δηλαδή πρόκειται ε, για τον μαύρο κατάλογο όπως είναι γνωστός. Εδώ έχουμε ένα, μια πρόταση ψηφίσματος από ε, τρεις εισηγητές. Ο κύριος Λουί Μισελ ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, βρίσκεται σε άλλη ε, ήπειρο. Αν δεν κάνω λάθος, δεν βλέπω ούτε καν τους άλλους, ούτε τους άλλους δύο εισηγητές. Okay. Mrs. Mrs. Mrs. Strifler is not here either because she's η κυρία Σνίφνερ βρίσκεται μαζί με τον κύριο Λουί ε, Μισελ και η κυρία Μποσκούρτ έρχεται. Ίσως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Λουί Μισελ και να υποβάλω ερωτήσεις στο Συμβουλίο αναμένοντας την ε, έλευση της κυρίας Μποσκούρτ για να μας κάνει μία εισήγηση και μετά το Συμβούλιο θα απαντήσει. Νομίζω ότι σε προγενέστερες ε, συναντήσεις έχουμε μιλήσει για τη νομική βάση και την απογοήτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι δεν συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία σε συνεργασία με το Συμβούλιο και αυτό είναι λυπηρό διότι το θέμα είναι ύψη της ε, σημασίας δεν αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αλλά και την ε, προστασία του κράτους δικαίου. Κατά το παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν ενδιαβουλεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με μέτρα για τη συναφή μέτρα για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Γι' αυτό μας εκπλήσει το γεγονός ότι δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία το Κοινοβούλιο. Επίσης, ποια νομική βάση χρειάζεται έτσι ώστε να έχουμε την ελάχιστη, τουλάχιστον, συμμετοχή, την ελάχιστη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά σε σχέση με τους μαύρους καταλόγους και είχαμε περιπτώσεις ε, του ΔΕΚ και εθνικές υποθέσεις σε σχέση με την ε, σύνταξη αυτών των μαύρων καταλόγων, την ε, ένταξη σημείων ή την αφαίρεση σημείων. Έχει επέλθει κάποια πρόοδος επί του θέματος. Αυτοί που εγγράφονται στον κατάλογο τουλάχιστον τους κοινοποιείται αυτό. Αυτή είναι και η βασική ιδέα, αλλά υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά για το πόση, πληροφορία, πόση πληροφόρηση έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που χρειάζονται και οι συνηγοροί τους έτσι ώστε να μπορέσουν να τους εκπροσωπήσουν. Υπάρχουν όμως και ε, άλλα σημαντικά ζητήματα, διότι αυτά τα μέτρα υποτίθεται ότι είναι προσωρινά. Τα πρόσωπα εντάσσονται προσωρινά, προληπτικά σε αυτούς τους καταλόγους, αλλά φαίνεται ότι ανά τον χρόνο ε, εντάσσονται μόνιμα, δηλαδή παραμένουν στον κατάλογο για μακρύ χρονικό διάστημα και η διαδικασία διαγραφής τους είναι περίπλοκη. Άρα έρεται ο προσωρινός χαρακτήρας των μέτρων. Επίσης θεωρείται διοικητικό μέτρο, αλλά αν τα φυσικά πρόσωπα παραμείνουν στους, μαύ, στους καταλόγους και αν δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τότε πρόκειται για μία ε, σαν δικαστική απόφαση και όχι προσωρινό μέτρο. Και θα ήθελα τέλος το Συμβούλιο να μας, πει ορισμένα, ε, να μας δώσει ορισμένα στοιχεία σε σχέση με την πολιτική φύση αυτής της διαδικασίας, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μία περίπτωση όπου η απόφαση του δικαστηρίου στην περίπτωση Σίσον μας έδειξε ότι πολλές φορές φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος, κίνδυνος έναντι της κοινωνίας ως προς την ε, ένταξη φυσικών προσώπων και πολλές φορές υπάρχουν και πολιτικά κίνητρα ένταξη στον κατάλογο. Παρά το γεγονός ε, ότι μιλώ αρκετή ώρα, βλέπω ότι η κυρία Μπόσκουρτ δεν έχει φτάσει ακόμα. Φαίνεται ότι είναι κάθοδον, αλλά πούντι. Τι θα κάνουμε θα περιμένουμε την κυρία Μπόσκορτ. Λοιπόν, περιμένουμε την έλευσή της. Στο μεταξύ το Συμβούλιο μπορεί να σκεφτεί τις απαντήσεις του. Um, Συνάδελφοι, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει ε, κάποιος από το Συμβούλιο, παρευρίσκεται κάποιος από το Συμβούλιο για να απαντήσει. Α, άρα μιλούσα μόνο στις κάμερες. Γιατί το Συμβούλιο δεν παρευρίσκεται, η εκπρόσωπο του Συμβουλίου, διότι δεν ε, υπήρχε αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Θα έπρεπε να είχαμε έναν ε, εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Κανείς δεν γνωρίζει το παραμικρό. Λοιπόν, ας διακόψουμε για 10 λεπτά και θα προσπαθήσουμε να βρούμε την εισηγήτρια και εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να καθίσετε σιγά σιγά, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Έχουμε και την εισηγήτρια εδώ, άρα σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Σίγουρα θα ζητήσει συγγνώμη επί μακρόν το Συμβούλιο ε, που μας τρώει το χρόνο. Αυτό πραγματικά είναι παράδεκτο. Okay, I see the Council has arrived, and I hope the rapporteur is not leaving the room now. Ήρθε η συγγήτρια, ήρθε και το Συμβούλιο, ελπίζω να μην φύγει η συγγήτρια τώρα. Κύριε Χάιντεν, καλώς ήρθατε. Περιμένουμε το Συμβούλιο κάπως η ώρα τώρα. Είχατε προβλεφθεί να είστε εδώ πριν από μισή ώρα. Μίλησα προσπαθώ, και αισθανόμουν τελείω ανόητη γιατί έκανα ερωτήσει προ το Συμβούλιο που δεν ήταν εδώ. Ε, πραγματικά είμαι δυσαρεστημένη. Τα ξαναλέω. Να καλέσω ωστόσο πρώτα τους, την κυρία Μποσκού, την άλλη συγκεκριμένη να κάνει την παρουσίασή τη. Παρακαλώ κύριε Μποσκούτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη για να δώσω την ευκαιρία και στους συναδέλφους που θα έρθουν και σε λίγο να πάρουν το λόγο. Στην παρούσα φάση έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος από τρεις ε, εισηγητές, Μισελ Στρίφλερ, Λουίς Μισελ και οι υποφαινόμενοι. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο για να συζητήσουμε τις γενικές γραμμές και τη διαδικασία. Δεν πρόκειται να επαναλάβω το περιεχόμενο του ψηφίσματος, το έχετε άλλωστε μπροστά σας, αλλά θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσει ότι θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να συμμετάσχει στην όλη αυτή τη διαδικασία και μιλάμε και μεταξύ άλλων και για άτομα τα οποία σχετίζονται με το δίκτυο της Αλκάιντα, το οποίο επηρεάζει και το ευρωπαϊκό δίκτυο. Μιλάμε για Ευρωπαίους πολίτες και όσοι εισηγητές θεωρούμε ότι είναι λογικό οι μελλοντικέ προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν διπλή νομική βάση και να έχουμε και δικαίωμα στην απόφαση εμείς στο Κοινοβούλιο. Υποβάλαμε το ερώτημα αυτό προ την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώ ω τώρα δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μα ε, έλθει αυτή η απάντηση. Περιμένουμε απάντηση, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην εβδομάδα. Τονίζουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί από ό,τι ξέρετε τα εμπλεκόμενα συμφέροντα είναι μεγάλα και είναι πολύ σημαντική η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά η αξιοπιστία της ε, διαδικασίας απαιτεί και την ενημέρωση του κόσμου, την ενημέρωση των κατηγορουμένων, προκειμένου να το γνωρίζουν ότι κατηγορούνται, να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Συμβουλίου, αναρωτιόμαστε αν όντως είναι αρκετά φιλόδοξες και αν ε, τηρούν και ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες και των συστάσεων του ΔΕΚ. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν το αίτημα αναθεώρησης και αξιολόγησης των μέτρων αυτών και τονίζουμε τη σημασία της προστασίας δεδομένων σε ό,τι αφορά και τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Μία συγκεκριμένη ερώτηση να απευθύνουμε προς το Συμβούλιο γιατί σήμερα είναι εορταστική ημέρα, εορταστική ατμόσφαιρα με την ε, εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Αναρωτιόμαστε αν ναι, το Συμβούλιο λοιπόν έχει λάβει, αν έχει λάβει η Επιτροπή μια συγκεκριμένη απόφαση, αν θα υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση και αν εμένει η Επιτροπή, αν επιμένει για να βασιστεί η όλη πρόταση επί του άρθρου 214. Αυτό το απευθύνω σε ερώτημα προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Μου είπαν ότι ο κύριος Μέλλε θα θα αντιπροσωπεύσει τον κύριο Στρίφλε. Θα ήθελα να σας πω ότι έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσα στα πλαίσια της διασφάλισης των ε, ελευθεριών. Ζούμε μία ειδική χρονική στιγμή και έχει μεγάλη σημασία να διασφαλίζουμε την ελευθερία σε όλες τις εκφάνσεις της. Και αυτό που έχει σημασία είναι να καταπολεμήσουμε πρωτίστως την ε, τρομοκρατία, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα όλου του κόσμου. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να λάβουμε υπόψη ότι η οποιαδήποτε τυχόν επίλυση του ζητήματος δεν θα πρέπει να είναι γραφειοκρατική υφή, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική ανάλογα με τις προσδοκίες των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό και το ΕΛΚ προωθεί αποτελεσματικά μέτρα για την πραγματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να επιτεθούμε κατά εκείνου που μας απειλεί και να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Λάβουμε υπόψη και την κλίμακα των αξιών μας πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις, τις εκφάνσεις, όπως είπα. Δηλαδή, αυτός ο οποίος πλήττει την ε, ανθρωπότητα πρέπει να τιμωρηθεί. Γι' αυτό θεωρούμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται πολύ σωστά. Ευχαριστώ κύριε Ντεμέλο. Η κυρία Μπόσκορτ επίσης αναφέρθηκε σε ορισμένα σημεία και θα ήθελα να πω εξ ονόματο των φιλελευθέρων ότι υποστηρίζουμε όλη την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, αλλά και το, το δίκαιο. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να προστατεύσει κανείς τους πολίτες κατά διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο να τους προστατεύει από τους τρομοκράτες. Και εάν ε, ληφθούν μέτρα κατά της τρομοκρατίας, να είδα ότι ζητήσατε το λόγο, Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά. Κάτι το οποίο δεν έγινε τα τελευταία χρόνια, διότι υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά για φυσικά πρόσωπα και φορείς που μπαίνουν στον μαύρο κατάλογο. Στην περίπτωση του κυρίου Σισόν ε, δεν ξέρουμε πώς ε, απείλησε την ασφάλεια των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και ε, ευτυχώς αθωώθηκε από τα δικαστήρια. Αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στην ένταξη, ως προς την ένταξη στον κατάλογο, στο μαύρο αυτό κατάλογο. Αποτελούν πραγματική απειλή. Γι' αυτό υπέβαλα και ερωτήματα στο Συμβουλίο ως προς την προσωρινή ένταξη στο μαύρο κατάλογο γιατί φαίνεται ότι πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο. Φαίνεται όμως ότι το μέτρο δεν είναι προσωρινό διότι όσοι εγγράφονται στη λίστα παραμένουν εκεί για μακρύ, χρονικό διάστημα. Και αυτό σχετίστηκε με το δεύτερο θέμα που έθιξα. Δηλαδή το Συμβούλιο μίλησε για τη διοικητική φύση του μέτρου αλλά επειδή πρόκειται για μόνιμο μέτρο είναι σαν να πρόκειται για μια δικαστική απόφαση. Τέλος, φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και πολιτική πίεση από ορισμένες χώρες που θεωρούν ότι τα φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις πρέπει να εγγραφούν στον κατάλογο για πολιτικούς λόγους και όχι για λόγους ασφαλείας. Θα θέλαμε το Συμβούλιο να απαντήσει, αλλά και ο κύριος Μπρόν ζήτησε το λόγο στο μεταξύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι εν πολλές, οι κατάλογοι είναι κενές μορφές ε, χειρονομιών, συμπεριφορών χειρονομίας. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Βλέπουμε περιπτώσεις όπου ο Σάμα Μπιν Λάντιν, η Αλ Καΐντα ε, δεν επιτυγχάνεται. Επιπλέον, οι Ταλιμπάν υπάρχουν σε δύο κατηγορίες. Καταρχά, κατηγορήθηκαν ότι παρέσχουν προστασία στον Οσάμπα Μπιν Λάντεν. Έκτοτε όμω, υπέστησαν μια σειρά πολέμου φθορά. Δεύτερον, υπάρχουν καθεστώτα μη δημοκρατικά, αλλά όχι κατά ανάγκη να απειλέ σε άλλες χώρε. Στην πρώτη κατηγορία, ο Σάμα Μπιν Λάντεν και η Αλκάιντα, θα ήταν πολύ καλό να έχουμε τον κατάλογο των μελών τους και να τον εντάξουμε στον κατάλογο, στη μαύρη λίστα. Δεν το έχουμε. Στην ουσία, είναι η οργάνωση ταυτίζεται με τα μέλη και είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τα συγκεκριμένα μέλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εμπλεκόμενοι στην λίστα ήταν πολίτες τρίτης γενιάς από το Πακιστάν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, Ε, μπαίνουν ε, σε υποπαραγωγούς ολόκληρες κοινότητες. Δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, να σταματήσουμε τη μετανάστευση από χώρε που παρέχουν τρομοκράτε και δεύτερον, να σταματήσουμε να κάνουμε πόλεμο στι μουσουλμανικέ χώρε που του οδηγεί σε δράση. Σε ό,τι αφορά του Ταλιμπάν, εγώ προσωπικά δεν του γουστάρω. Δεν θα ήθελα να μένω υπό, να ζω υπό κυβέρνηση Ταλιμπάν και πολλοί άλλοι το ίδιο. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να διεξάγουμε ένα φρικτό πόλεμο κατά του Αφγανιστάν συνολικά για να ανατρέψουμε μια κυβέρνηση, προγενέστερη κυβέρνηση μάλιστα που δεν μας αρέσει, δεν είναι η δουλειά μας. Σε ό,τι αφορά γενικά τα καταπιεστικά καθεστώτα τη Ζιμπάμπου για παράδειγμα, νομίζω ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να προστατεύουν τα συμφέροντα των πολιτών τους που υποφέρουν από αυτή την ε, καταστολή και να καταδικάζουν τα συστήματα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάει να βάζουμε την κυβέρνηση των ε, ε την της κυβέρνησης της Ζιμπάμπου στον κατάλογο. Επιπλέον, ε, βασική γραμμή νομίζω στο κείμενο είναι να μην παραδώσουμε ποτέ και επαναλαμβάνω ποτέ άτομα σε χώρες δημοκρατικά ή όχι που επιβάλλουν στα άτομα αυτά την έκτακτη παράδοση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάτφορντ και μετά η κυρία Φλότορ. Νομίζω ότι Καλό είναι αυτό το, η όλη δουλειά που κάνουμε στην έκτακτη παράδοση. Ιδίω δε στην αιτιολογική σκέψη Γ που αναφέρεται στο ότι τα στοιχεία που υπάρχουν για να αποδείξουμε την επιτυχία του καθεστώτος αυτού θα πρέπει να μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε όχι μόνο την επιτυχία των κυρώσεων αλλά και το ότι η Επιτροπή αυτή είναι, δείχνει την επιτυχία ενός καθεστώτος που αποφασίζει την διακοπή τρομοκρατικών πράξεων και εγκλημάτων. Φαίνεται ότι τα μέτρα και η οδηγία για την, το ξέπλυμα του χρήματος και την χρηματοδότηση των ε, τρομοκρατών. Πλήττει στην πράξη πολίτε που προσπαθούν να απλού πολίτε στη χώρα μου τουλάχιστον που προσπαθούν να ανοίξουν λογαριασμό, αλλά δεν μειώνουν την σφαγή και τους βιασμούς σε χώρε όπως το Κονγκό. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε συνολικά το πού θέλουμε να πάμε. Το είπα και εσείς πρόεδρε για το καθεστώς PNR χρειάζεται πάντα να έχουμε σαφή εικόνα της χρησιμότητας των μέτρων. Δεν λέω ότι δεν είναι ποτέ απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε αυτά τα έκτακτα μέτρα ή υπομορφή προσωρινών περιορισμών, αλλά ανα πάσα περίπτωση και ανα πάσα στιγμή θα πρέπει να προχωρούμε προς την κατεύθυνση της άγκληση αποδεικτικών στοιχείων για να δικάσουμε τα συγκεκριμένα άτομα, ούτως ώστε να έχουν μια δίκη δίκη με τα απαραίτητα χέγγια. Αυτά τα γκρίζα καθεστώτα δεν είναι ικανοποιητικά σε σχέση με την εφαρμογή διαδικασιών ποινικού δικαίου. Η κυρία Ευχαριστώ. Να σας πω ότι καταρχάς η έκθεση είναι πολύ καλή, το θέμα, ενώ το θέμα είναι δύσκολο. Η νομική υποστήριξη για την επέκταση του δικαιώματος διαβούλευσης και των βάσεων νομίζω ότι είναι θεμελιωμένο. Μέσα στο πνεύμα της Λισαβόνας μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις θέσεις του Συμβουλίου σχετικά. Εγώ προτείνω, επειδή η έκθεση μιλά για την ανάγκη να υπάρξουν benchmarks στο σύστημα των κυρώσεων, αναγκαίο κατά την άποψή μου, για να μπορέσουμε να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων αυτών, όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε. Πρόκειται πάντα για πολύ δύσχριστά μέσα και η κυρώσει είναι και ένα πολιτικό εργαλείο. Γι' αυτό σε μια έκθεση πρωτοβουλία πριν την προηγούμενη θητή είχαμε ψηφίσει υπέρ τη δημιουργία ενό δικτύου ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων που θα είχαν στόχο να συνοδεύουν την Επιτροπή σε αυτό το δύσκολο έργο. Και νομίζω ότι μπορούμε χρήσιμα στην έκθεση αυτή, αν μου το επιτρέψουν οι ΣΥΤΕΣ, να το πω να προσθέσουμε την πρόταση αυτή στην έκθεση, θέση που είναι ήδη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατόπιν, στην παράγραφο 10 μιλάτε για την ανάγκη το Εθνικό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν την ικανότητα αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των, υπηρεσιών, των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ε, αντικατασκοπίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι αναγκαίο Νομίζω ότι είχαμε υποστηρίξει και ψηφίσει πριν από λίγο καιρό την ιδέα να μετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, διάσκεψη των υπηρεσιών παρακολούθησης των υπηρεσιών πληροφόρησης των κρατών μελών. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να το ξαναπούμε. Χρήσιμο θα είναι και ε, επί του πρακτέου. Κύριε Μέλο, Ζητήστε ξανά το λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Μετά από την ε, δική σας παρέμβαση θα ήθελα και πάλι να λάβω το λόγο. Συμφωνώ με αυτά που είπατε, ε, Πρόεδρε, αλλά πιστεύω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα των δημοκρατικών καθεστώτων έγκυται στο γεγονός ότι ότι τηρούν διαδικαστικά οτιδήποτε έχει σχέση με την εγγύηση των ελευθεριών. Αλλά ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αυτό το μεγαλείο της δημοκρατίας του αφαιρεί την αποτελεσματικότητα ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δηλαδή, για λόγους κοσμιότητας θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο επιθετικοί στην καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποιος επιλέγει την τρομοκρατία ως τρόπο ζωής και στόχο ζωής δεν έχει, δεν προβάλλει μία αντίρροπη δύναμη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που στο αστικό δίκαιο μιλάμε, ε, αναφέρουμε ως ρήξη δικαιωμάτων. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι ανάμεσα στα δύο δικαιώματα να δούμε ποιο υπερέχει. Αφενός, λοιπόν, θέλουμε να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα στην καταπολέμηση της δημοκρατίας, αλλά μιλάμε και για την επικύρωση των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ε, σεβόμαστε και να τηρούμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του πολιτή. Τη στιγμή όμως που υπάρχει ρήξη συμφερόντων και δικαιωμάτων θα πρέπει να δούμε κατά πόσο δεν πρέπει να καταστήλουμε δικτατορικά καθεστώτα όπως αυτό της Ζιμπάμπουε και της ε, Σομαλίας. Έχω όμως μία επιφύλαξη. Όταν μιλάμε για τρομοκρατία, μιλάμε για μία δραστηριότητα που πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όταν μιλάμε για μία χώρα όπως τη Ζιμπάμπουε, λαμβάνουμε υπόψη ένα καθεστώς που παρά τα αρνητικά του χαρακτηριστικά δεν πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Την πλήττει μόνο αν ε, ε υποθάλπει εγκληματίες και ε, τρομοκράτες. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την διασφάλιση αυτών των ελευθεριών ως προς ε, δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών θα πρέπει να μιλάμε για συνολική υπεράσπιση, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι μια υποχρέωση που μας αφορά όλους. Θα πρέπει όμως επίσης να γνωρίζουμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε να κάνουμε με τρομοκράτες και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με ελεύθερους πολίτες που θέλουν να παραμείνουν ελεύθεροι και δεν θέλουν να πλήτεται η καθημερινή του ζωή επειδή υπάρχει τρομοκρατία. Ε, σας κατανοώ απόλυτα, αλλά ήθελα να μιλήσω για αυτή την κλίμακα αξιών. Διότι πολλές, σε πολλές περιπτώσεις τα όπλα, το πλωστάσιο δεν είναι το ίδιο. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξέρουμε τι περιλαμβάνει αυτή η προστασία γιατί διαφορετικά το κόστος μπορεί να είναι η ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, δεν έρχομαι σε αντίθεση με αυτά που είπατε, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να προσαυξήσω ε, τη δήλωσή σας. Ευχαριστούμε. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, ε, κύριε Μέλο, όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των εγκληματικών καθεστώτων. Δεν συμφωνώ μαζί σας ως προς το εξής. Πολλές φορές γίνεται λόγος για εθνική ασφάλεια για να προσπίσουμε αυτά τα δικαιώματα και αυτό δεν οδήγησε σε μεγαλύτερη ασφάλεια των πολιτών. Και πιστεύω ότι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές δοκιμάζουμε τα συστήματά μας, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων. Θα ήθελα το Συμβούλιο να σχολιάσει και να απαντήσει. Η κυρία Χάιντινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησα ως προς την έλευσή μου. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ μαζί σας θα πρέπει να προωθήσουμε μέτρα αντιμετώπισης ε, της τρομοκρατίας, αναχέτησης της τρομοκρατίας και θα πρέπει να προωθήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων που πλήττονται με αυτά τα μέτρα. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να σας απαντήσω και θα μου πείτε κατά πόσο ε, αν και κατά πόσο δεν τα καταφέρνω καλά. Νωρίτερα τον Νοέμβριο σας είπα και επαναλαμβάνω ότι οι κυρώσεις αποτελούν ένα στοιχείο της πολιτικής μέσα στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας να βελτιώσουμε την κατάσταση σε τρίτες χώρες. Οι κυρώσεις δεν είναι η μαγική φόρμουλα η οποία θα καταστήλει τις βίες πράξεις μιας ε, κατασταλτικής κυβέρνησης και οι κυρώσεις δεν αποκλείουν και άλλες δραστηριότητες που θα πρέπει να συνεπάρχουν όπως αναπτυξιακές δραστηριότητες, διάλογος με μη κυβερνητικές και ούτω καθεξής. Ίσως ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δραστηριότητες πρωτίστως με τις μη κυβερνητικέ. Άρα οι κυρώσεις δεν είναι το μόνο μέσον για την βελτίωση της θέσης μιας χώρας. Όταν όμως εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η απαγόρευση, η απαγόρευση χορήγησης θεώρησης θα δεν θα επιτρέψει στους ε, επικεφαλείς κυβερνήσεων να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη ενώ οι λαοί τους ε, λιμοκτονούν. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να δούμε το συγκριτικό πλεονέκτημα ορισμένων μέτρων και ως προς τον ε, αποκλεισμό, αποκλεισμό διακίνησης όπλων δεν θα επιτραπεί η πώληση όπλων από την Ευρώπη σε αυτές τις χώρες. Μπορούμε λοιπόν να εισαγάγουμε μέτρα που να σχετίζονται με τις δικές μας δραστηριότητες. Δεν έχουμε ε, επιπλέον εδαφική δικαιοδοσία. Γι' αυτό οποιαδήποτε μέτρα αποφασίσει να εφαρμόσει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ισχύσουν σε εμά. Και αυτό αποτελεί μια εγγενή αδυναμία των κυρώσεων αν δεν αποφασιστούν σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, διότι τότε θα υπάρχει παγκόσμιος αντίκτυπος. Αλλά και εμείς θα πρέπει να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι έτσι ώστε να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα ήταν ε, σκόπιμο να πω ότι από πλευράς ε, τρομοκρατίας έχουμε διαφορετικούς τύπους μέτρων. Αφενός μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και που σχετίζονται με το ψήφισμα 1267 των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τον κανονισμό 881 που ονομάζουμε κανονισμό Ταλιμπάν, ο οποίος τώρα αναδιατυπώνεται και γνωρίζεται το περιεχόμενο αυτού του κανονισμού. Ακριβώς εδώ προτείνουμε να εντάξουμε ε, επιπρόσθετες ρήτρες διασφάλισης σε σχέση με αυτά που μας είπε το ΔΕΚ στην απόφαση του, του παρελθόντος Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα μέτρα που αποφάσισαν και τα Ηνωμένα Έθνη, διότι είπαμε ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των αποφάσεων του ΔΕΚ και όπως τονίσατε και στο δικό σας ψήφισμα, δηλαδή μέτρα που προωθεί το, ε, τα Ηνωμένα Έθνη στα πλαίσια του ψηφίματος 18-22. Επίσης υπάρχουν και ανεξάρτητα μέτρα τα οποία βασίζονται στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά όπου το ε, Συμβούλιο αποφασίζει ως προς ανεξάρτητους καταλόγους και εμείς θα πρέπει να αναθεωρούμε το όλο πλαίσιο αναεξάμεινο ως προς τους ε, καταλόγους αυτούς που ισχύουν σε συνεχή βάση, δηλαδή να γίνεται μια εξαμηνιαία αναθεώρηση και σε αυτά τα πλαίσια τα φυσικά πρόσωπα, οι οντότητες ε, την χάνουν αναθεώρησης. Σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία, νομίζω ότι μία ε, μεγάλη βελτίωση, όπως τόνισε και το ΔΕΚ, είναι το το καθήκον τεκμηρίωσης ε, για την εγγραφή στο μαύρο κατάλογο φυσικών προσώπων ή οντοτήτων. Και ακριβώς αυτό κάνουμε. Ως προς την φύση αυτών των μέτρων, δεν είναι ε, δικαστικού χαρακτήρα, δικαιοδοτικού χαρακτήρα, διότι το Συμβούλιο δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο. Είναι πολιτικές και μέτρα τα οποία πάντα λαμβάνουν υπόψη τις νομικές ρήτρες ε, διασφάλισης. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνουμε δεν θα πρέπει να είναι γραφειοκρατική η φύση η χαρακτήρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι πιστεύουν οι συνάδελφοι, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι μία απάντηση δεν απαντήθηκε. Συμφωνήσατε ότι παρουσιάστηκε αυτό ως προσωρινό διοικητικό μέτρο. Το γεγονό όμως ότι φαίνεται ότι κάποια άτομα παραμένουν επί σειρά ετών στον κατάλογο αυτό, αφαιρεί καταλαβαίνετε το προσωρινό του μέτρου αυτού. Πρόκειται για δικαστική απόφαση. Και το δεύτερο θέμα που ήθελα να θίξω είναι το εξή. Στην εισαγωγή σα φαίνεται να αναφέρετε από κοινού κάποια μέτρα, για παράδειγμα κατά των ε, ηγετών της Σιμπάμπουε, όπου φυσικά όλοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε για εδώ ή για παράδειγμα υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις του Συμβουλίου αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο, θεωρώ, με το να βάζουμε οργανώσεις ε, στο κατάλογο για να στερήσουμε την ροή χρημάτων σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Στη μία περίπτωση μιλάμε για πολιτική δράση υπέρ του εκδρομοκρατισμού, για παράδειγμα της Ιμπάμπουε. Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για θέμα ασφάλειας, όπως είπε και ο κ. Μπρόντς είναι λίγο, είναι δύο τελείως διαφορετικά είδη μέτρων. Συνάδελφοι, δεν ξέρω, σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις που λάβατε. Ωραία. Ο κύριος Μπρόνς και η κυρία Μποσκούρτ. Να ακούσουμε τι έχετε να πείτε κι εσείς και μετά να επανέλθουμε στο Συμβούλιο. Ναι, μπορεί να μου διέφυγε αλλά δεν θεωρώ ότι διασαφηνίστηκε η ερώτηση που έθεσα προς το Συμβούλιο για το κατά πόσο έχει ληφθεί ή όχι οριστική απόφαση υπό το παλαιό καθεστώς και κατά πόσο θα ακολουθήσει νέα πρόταση. Δεν ξέρω, μπορεί να μην κατάλαβα και εγώ. Θα ήθελα όμως να έχω μια σαφή απάντηση. Και επί της νομικής βάσης επίσης. Κύριε Μπρόντς. Uh, Ευχαριστώ. Είναι πολύ μικρό το θέμα αυτό που ήθελα να θίξω. Το εξή. Φαίνεται ότι μας αναστατώνουν χώρε όπως η Ζιμπάμπουε, οι οποίες όμως είναι σχετικά αδύναμες. Όταν μιλάμε για μεγάλους καταπιεστές όπως η Κίνα, που δεν καταπιέζει μόνο το λαό τη, αλλά και εκτελεί πολύ κόσμο για σχετικά μικρά αδικήματα, σιωπούμε. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα πρότυπο θα πρέπει να το εφαρμόσουμε με τον ίδιο τρόπο σε όλους, μάλιστα. Αυτό ακούγεται πολύ επαναστατικό σε σχέση με την παράδοσή μας. Ο κύριος Μέλο και μετά το Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μπρόνς ότι συμφωνώ απόλυτα δεν νομίζω ότι σε αυτή την αξιολόγηση που γίνεται για το κράτος της Ζιμπάμπουε μπορούμε να ξεχάσουμε το γεγονός ότι στη ε, Ζιμπάμπουε πολλές φορές ε, γίνονται εγκλήματα χωρίς να ε, έχει διαπράξει το φυσικό πρόσωπο κανένα ούτε καν τέσμα πολλό δε μάλλον πλημέλημα. Πολλές φορές δεν έχει διαπράξει τίποτα. Απλώς προβάλλει το δικαίωμα λόγου και σε, στην περίπτωση της Κίνας δεν μπορούμε παρά να σχετικοποιήσουμε ε, ως προς το τι συμβαίνει στη Ζιμπάμπουε. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Κίνα ή στο Ζιμπάμπουε, οπουδήποτε στον κόσμο, δεν μπορώ να δεχτώ οποιοδήποτε ε, καθεστώς να μην επιτρέπει την ελευθερία λόγου στους κατοίκους του, δηλαδή να φυλακίζει τα πρόσωπα αυτά και να τα σκοτώνει. Δηλαδή αυτό που ισχύει και στην Κίνα και στο Ζιμπάμπου είναι απαράδεκτο. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρισκόμαστε στην πλευρά του νόμου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, προσπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη από τη Ζιμπάμπουε στην Κίνα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την, ε, τα κατασταλτικά αυτά καθεστώτα κατά ε, ανθρώπων, μικρών παιδιών, γυναικών, αθώων δεν μπορούμε να δεχτούμε την περιστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Απλώς τα όπλα δεν είναι τα ίδια. Βεβαίως υπάρχουν κατάλογοι που, όπου ένα πρόσωπο στιγματίζεται διότι η περίπτωσή του δεν επιλύεται δικαστικά. Όμως υπάρχουν πολλές χώρες όπου στη δική μου χώρα, όπου κανείς είναι κατηγορούμενος για ε, χρόνια, γιατί το κράτος ε, δεν μπορεί να απαντήσει σε σχέση με τραπεζικές ε, πρακτικές, με θέσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με, δημόσια, με θέματα δημόσιας διοίκησης και ούτω καθεξής. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε πολλές φορές με συγχωρείτε, πρέπει να σας διακόψω, γιατί βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων προς το Συμβούλιο. Έχετε μια ερώτηση προς το, ε, προς το Συμβούλιο. Ναι, ε, την ίδια ερώτηση με τον ε, προλαλήσαντα. Okay, thank you. So Το ερώτημα για την νομική βάση και την ερώτηση για την συνοχή της προσέγγισης γιατί κάποιες χώρες και όχι άλλες. Αλλά υπάρχει και ερώτηση σχετικά με τον προσωρινό και διοικητικό χαρακτήρα των μέτρων και πώς μπορείτε να, δια... Ε, βεβαιώσετε ότι κάτι θα ισχύει ενώ ο κόσμος είναι στους καταλόγους αυτούς ε, σχεδόν εσαΐ. Ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Πρώτο θέμα. Νομική βάση. Όπως ξέρετε, το Συμβούλιο υπέβαλε τον κανονισμό 881 για το ΕΣΕΛΟΝ, ζητώντας τη γνωμοδότησή σας παρά τη νέα συνθήκη και όπως ξέρετε δεν, δεν υιοθετήσαμε την απόφαση του Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε την ε, απόφαση του Κοινοβουλίου για να τη λάβουμε υπόψη πριν εγκρίνουμε τον κανονισμό. Έτσι θα προχωρήσουμε στο ζήτημα αυτό. Χρηματοδότηση δημοκρατικών δραστηριοτήτων και συνοχή. Αυτές είναι αποφάσεις πολιτικής που συζητώνται βεβαίως. Για κάποιες χώρες ή για κάποια θέματα, το είπα και στο ξεκίνημα, μέτρα που λαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν την τάση να είναι πιο αποτελεσματικά από μέτρα που υιοθετούνται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εκ των πραγμάτων έχουν περιορισμένη εμβέλεια μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου να θεωρηθεί σημαντικό πολιτικά να επιβάλλονται μέτρα για να βοηθηθεί μία συγκεκριμένη χώρα ή για να επιτρέψουμε σε μία συγκεκριμένη χώρα να αλλάξει τις πολιτικές της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προσωρινό χαρακτήρα των, μέτρων, των διοικητικών αυτών μέτρων, να σας πω, είναι, ναι, είναι διοικητικά μέτρα που βασίζονται στις εθνικές αρμόδιες ε, αρχές δικαστικού χαρακτήρα. και βασίζονται σε νόμιμες αποφάσεις για το πάγωμα κάποιων περιουσιακών στοιχείων, για παράδειγμα. Να υπογραμμίσω επίσης ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχουν αυτές οι αναεξάμεινο αναθεωρήσεις και ότι πραγματοποιούνται. Και άρα υπάρχει μια βεβαίωση ότι κάθε έξι μήνες θα λαμβάνεται μια απόφαση για το κατά πόσον άτομα ή φορείς που εντάσσονται στον κατάλογο αυτό θα μείνουν ή όχι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των Ταλιμπάν και της Αλκάιδα, παίρνουμε την απόφαση, ακούμε τις απόψεις και μετά την παρουσίαση των απόψεων λαμβάνουμε τη δική μας απόφαση. Οι αναθεωρήσεις που κάναμε με βάση τον αυτόνομο κατάλογο οδήγησε στο να βγουν περί τα 20 άτομα από τον κατάλογο και 6 ομάδες από το 2002 και μετά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για τις τροπολογίε στο ψήφισμα, για το ψήφισμα αυτό είναι 3 Δεκεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου, την άλλη Δευτέρα. Κατόπιν υποθέτω ότι προβλέπεται να εγκριθεί στην Ολομέλεια αυτού του Στρασβούργου. Ωραία, ευχαριστώ. Τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η δημιουργία αξιωματικών ενός δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. Θα ακούσουμε τον εισηγητή, την εισηγήτρια κυρία Τον εισηγητή κύριο Ντίας συγγνώμη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, η έκθεση αυτή Είναι τρίτη φορά που την εξετάζουμε και τη σχολιάζουμε στην Επιτροπή μας. Προέκυψαν κάποια καινούργια στοιχεία που καλό θα ήταν να γνωρίζετε. Κάποια από τις αλλαγές τις έμαθα εγώ πριν από μισή ώρα, ούτε καν μισή ώρα, χάρη στην πολύ καλή δουλειά του Εμίλιο Τεκαπιτάνη που με ενημέρωσε. Πρώτον, να ευχαριστήσω ιδίω τους συναδέλφους για τις τροπολογίε που υπέβαλαν στην έκθεση. Την κυρία Ηλιόμ 8, την κυρία Βίξτον 5, την κυρία Κίλε 4 και Φλότο Κίλε με άλλους 3, Μοθού 2 και, Ρίτα, και, κύριο, και ο κύριος Ταβάρης 2. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί όλες οι τρομολογίες με βοηθούν και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την έκθεση. Δεύτερον, έχουμε χρόνο κάποιες τροπολογίες που αφορούν με την ορολογία που χρησιμοποιούμε για να διακρίνουμε την όρου λάθρο μετανάστευση, παράνομη μετανάστευση, ε, κακός, μη τακτοποιημένη μετανάστευση είναι ένα ζήτημα που το προσπάθησα να το καλύψω και εγώ για να μην δημιουργούμε ατυχείς, ε, Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιούμε τον όρο ε, irregular ή clandestine και όχι το illegal, όχι το παράνομο, αλλά το λάθρο ή το μη τακτικό. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάποιες χώρες ο όρος παράνομος είναι όρος του ποινικού δικαίου. Άρα κάποια κράτη μπορούν να δεχθούν τη διαγραφή του όρου παράνομος, αλλά άλλα κράτη θα μας κατηγορούσαν ότι μπαίναμε σε εθνικά εδάφη αν καταργούσαμε τον όλο παράνομος. Εγώ λοιπόν προτείνω τον όρο clandestine που στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως λάθρο μετανάστευση. Έναν όρο που μπορούμε να συνοψίσουμε και να αποδεχθούμε από τις εμπλεκόμενες, τις διαφωνούσες πλευρές. Εγώ πάντως σας δηλώνω εξ αρχή ότι δεν θέλω να μιλήσω για παράνομη μετανάστευση. Ίσως λοιπόν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε τον όρο clandestine ή irregular. Άλλα ζητήματα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω ή δεν μπορώ να δεχθώ ή για προφανείς λόγους. Συνήθως είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του κανονισμού που θέλουμε να αλλάξουμε. Θα κάνω κάποια σχόλια για τις προτάσεις αυτές προσπαθώντας να πετύχουμε συνένεση στις υπόλοιπες γιατί έχουμε ένα ζήτημα στην απόφαση. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να έχουμε μεγάλη συνένεση νέο στοιχείο που είπα και για το οποίο με ενημέρωσε ο Εμίλιο προηγουμένω ήταν ένα θέμα που εξέτασα τελείω επιφανειακά γιατί δεν είχα χρόνο να το δω στη μισή ώρα που είχα στη διάθεσή μου, αλλά που δεν μου κακοφαίνεται και δέχομαι καταρχήν. Η Επιτροπή προτείνει αλλαγή τη νομική βάση. Θα θυμάστε ότι η νομική βάση που μα είχε υποβληθεί ήταν το 63-3-Β και το 66 της συνθήκης. Η Επιτροπή τώρα προτείνει να αλλάξει νομική βάση ως εξής. Προτείνει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 74 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλά για τη διοικητική συνεργασία και την χρήση του άρθρου 79 για τη μεταναστευτική πολιτική και ως στόχο την παράγραφο 2 γάμα που αναφέρεται στην λάθρο μετανάστευση και παράνομη, μη, μη ε, νόμιμη ε, διαμονή. Clandestine και irregular χρησιμοποιεί στο κείμενο. Τι συμβαίνει με τη Λισαβόνα τώρα. Με τη Λισαβόνα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα την νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή εισάγοντας το άρθρο 71α μικρό που μιλά για νόμιμη μετανάστευση, ένα βασικό κομμάτι της έκθεσης και την μακράς διάρκειας νόμιμη μετανάστευση. Θα μπορούσαμε λοιπόν καταρχήν να συμφωνήσουμε με την εισαγωγή του άρθρου 74α. Τρόπος λειτουργίας. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Οπότε θα μπορούσαμε να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή και ταυτόχρονα να ξεκινήσουμε πιο ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις με τους ε, συντάκτες των απολογιών για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση. Αυτά και ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει κάποιος να σχολιάσει ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ. Εντάχει, σε σχέση με την ορολογία, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να προωθήσουμε θέματα ε, ορολογίας θα ήταν να οριοθετήσουμε καλύτερα τους όρους, αλλά στο αφήσουμε κατά το ζήτημα, κατά μέρος τώρα το ζήτημα από γλωσσικής, γλωσσολογικής πλευράς. Αυτό που έχει σημασία είναι να βελτιώσουμε τη δική μας κατάσταση δέχομαι αυτά που είπε ο κύριος Δίας Δεμέρα ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μία συμφωνία επί των όρων. Δηλαδή ο όρος ε, η regular είναι πιο περιοριστικός. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ευρύτερο όρο έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για να δούμε κατά πόσο καλύπτουμε αυτή την πραγματικότητα και αυτό αφορά την ε, λαθρομετανάστευση, την ε, παράνομη μετανάστευση. Γι' αυτό νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να μιλάμε για irregular Η illegal είναι παράνομος καθαρά, αλλά δεν είναι σωστός ο όρος αυτός. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ε, εξεύρουμε μία λύση που να μας βρίσκει ε, σύμφωνους όλους σε σχέση με το irregular και το clandestine. Αλλά νομίζω τελικά ότι το illegal δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τώρα, σε σχέση με άλλες τροπολογίες ε, που υπέβαλα, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα, διότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όταν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον φορέα αυτό. Τη στιγμή που μιλούσαμε μέχρι τώρα για το Frontex, το ΕΑΣΟ δεν υφίσταται ακόμα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να σκεφτεί ακριβώς πώς θα αντιμετωπίσει και το θέμα των προσφύγων. Δηλαδή θα πρόκειται για έναν κεντρικό φορέα πώς θα διαχειριστούμε αυτό το ΕΑΣΟ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για θέματα ασύλου. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές. Ελπίζω να υπάρξει συνένεση έτσι ώστε οι αξιωματικοί σύνδεσμοι να έρχονται συνεχώς σε επαφή και με το Frontex και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρη. Ο επόμενος, η επόμενη μάλλον η κυρία Κέλλερ και μετά η κυρία Γκίου. Ευχαριστώ. Οι τροπολογίε μας ουσιαστικά κινούνται προ δύο κατευθύνσει. Καταρχάς, ότι θέλουμε να υπάρχει πιο καλή ενημέρωση του Κοινοβουλίου για να ξέρουμε ποιε εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια είναι τα αποτελέσματά του. Γιατί αυτό δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση. Κατά δεύτερον, θεωρούμε ότι αν αυτοί οι αξιωματικοί σύνδεσμοι για την ε, μετανάστευση πρέπει να συνεργάζονται με τις χώρες, είναι σημαντικό να εξετάζουν πώς έχει η κατάσταση σε κάθε χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι κάνει η κυβέρνηση, τι, κάνει, τι κάνουν οι αρχές με τους πρόσφυγες και για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιο μεταναστευτικό ρεύμα. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν αν θέλουμε όντω να καταπολεμήσουμε τα θέματα τη λαθρομετανάστευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κιού. Ε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις απόψεις που εκφράστηκαν ότι δεν μπορούμε να, να αποφασίσουμε επί του θέματος αυτού οριστικά τώρα. Πιστεύω ωστόσο ότι χρειάζεται να γίνει λίγη ακόμα δουλειά για να συμφωνήσουμε ως προς την ορολογία. Αν το λάθρα ταιριάζει σε όλες τις ε, περιπτώσεις και στο κείμενο εν γέννη. Ίσως χρειάζεται λοιπόν και άλλη δουλειά. Δεύτερο θέμα. Τρία μάλλον έχω συνολικά. Το δεύτερο άσυλο. Άκουσα τι έλεγε ο κύριος Σταβάρης για την επαφή με το γραφείο και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος για το περιθώριο δουλειάς του δικτύου με το γραφείο αυτό, ούτως ώστε, και αυτό είναι, αυτό είναι το τρίτο μου σημείο, έτσι ώστε ο ρόλο που θα ανατεθεί στο μέλλον στους στο δίκτυο αυτό αξιωματικών συνδέσμων να μην γίνει υπερβολικά ασαφής. Ε, υπάρχει μια τάση που διαβλέπω να προσπαθούν να τους δώσουν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, να κάνουν τα πάντα και να μην έχουν κάτι συγκεκριμένο, ένα συγκεκριμένο στόχο. Να τονίσω και κάτι ακόμα. Το κείμενο αναφέρει ότι οι αξιωματικοί σύνδεσμοι υποβάλλουν αναεξάμεινο εκθέσει στο Συμβούλιο. Να σας πω ότι στις 9 Νοεμβρίου ζήτησα να δω τις τελε... τρεις τελευταίες εξαμηνιαίες εκθέσεις. Δεν έλαβα ακόμα οποιαδήποτε απάντηση από οποιονδήποτε για το θέμα αυτό. Είμαι υπομονετική βέβαια, περιμένω, αλλά αν θέλουμε να εμφανίζονται, να ετοιμάζονται και να ανακοινώνονται κατόπιν οι εκθέσεις αυτές στο Κοινοβούλιο, κάπως πρέπει να το δούμε. Σίγουρα είναι προσωρινό προβληματάκι. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ. Η ιδέα να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων για τη γλώσσα, για τους όρους που θα χρησιμοποιούμε είναι περιοριστικό. Και ο Όργουελ έλεγε ότι όσοι περιορίζουν τη γλώσσα περιορίζουν τη σκέψη και τη συζήτηση. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει μια διατύπωση που θα περιλάμβανε τον όρο μετανάστευση, που είναι παράνομη ή όχι, χωρίς άδεια, μια εγκεκριμένη δηλαδή, αλλά τέλος πάντων αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι να επιλέξει ο καθένας την έκφραση στη γλώσσα που ε, εκφράζει καλύτερα τις ε, θέσεις και τις ε, παραδοχές. Κάποιο είπε το πρωί, και δεν είναι λάθο, ότι δεν πρέπει να κάνουμε ιδεολογικέ μάχε, να τι αφήσουμε κατά μέρο. Μπράβο. Αυτό πολύ σωστό. Και νομίζω ότι πρέπει να το εφαρμόσουμε παντού. Ευχαριστώ κύριε Μπροντ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει το λόγο. Δίνω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή εκ νέου. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ακριβολογήσω σε σχέση με αυτό που παρέμεινε ανοιχτό για περαιτέρω διευκνήσεις που ε, χρησιμοποιώ ορθολογικά. Σας είπα ότι μέσα στα πλαίσια του κόμματός μου και εκτός θεωρώ ότι θα πρέπει να διαγράψουμε το illegal, το παράνομο. Τώρα όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν πρόκειται για σημασιολογικό θέμα. Είναι και σημασιολογικό και νομικό. Και επειδή ακολουθούμε αυτή την σειρά, δηλαδή νομικό και σημασιολογικό, θα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση η οποία να μην πλήττει τις εθνικές νομοθεσίες. Γι' αυτό, συμφωνώντας ε, καταρχήν με την ε, αρχή Α, θεωρώ ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε το ε, δεύτερο σκέλος. Τώρα, σε σχέση με τη, τη λέξη παράνομος, κλαντεστίνο, επειδή μιλάμε για καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και επειδή θεωρώ ότι οι μεταναστευτικές ροές δημιουργούν μεγάλα ευεργετήματα και για τις χώρες υποδοχής και για τις χώρες προέλευσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα έτσι ώστε για να φτάσουμε σε μία συνένεση να έχουμε και νομική κάλυψη και σημασιολογική κάλυψη στους όρους που, ως προς τους όρους που χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι αυτό δίνει μία απάντηση στα σχόλια του κυρίου Ταβάρες, της κυρίας Γιουγιόμ και του κυρίου Μπρόνς. Τώρα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, εγώ δεν αντιτίθεμαι έτσι ώστε η υπηρεσία αυτή να αποτελέσει μέρος του πουλ ε, Frontex και ε, αξιωματική σύνδεσμη. Αυτό μας τι σημαίνει. Θα σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο για να υπάρχει αυτή η ομαδοποίηση, αυτό το pooling και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους απότερους στόχους που είναι τέσσερις ως προς την πρόταση τροποποίησης. Δεν θα σας διαβάσω την πρόταση για να μην μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να την διαβάσετε την πρόταση. Εγώ δεν αντιτίθεμαι καταρχήν να, να συμμετάσχουμε στην υπηρεσία για θέματα ασύλου. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ καταπολέμησα τις ε, καθυστερήσεις, τις αναβολές και θεώρησα το Ταμείο για τους πρόσφυγες που είναι 628 εκατομμύρια ευρώ έδωσα μάχη έτσι ώστε το Ταμείο Προσφύγων να μην χρησιμοποιηθούν μάλλον χρήματα από το Ταμείο των Προσφύγων για να δημιουργηθεί η Άσο. Τώρα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση περιλαμβάνει μία μνήα στα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες προέλευσης. Αυτό μας είπε και η κυρία Χίλερ. Αυτό ήδη γίνεται. Αλλά καλό να το θέσουμε και επί χάρτου. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ποιότητα τήρησης των ανθρωπίνων και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες προέλευσης που δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Η κυρία Γκυγιόμ αναφέρθηκε στις εξαμηνιές εκθέσεις. Μακάρι να υπάρχει γρήγορη πληροφόρηση σε αυτό που θέλετε, αλλά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μπάς περιπτώσει, δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εξαμηνιαίων εκθέσεων. Υπήρχε μεγάλη διχογνωμία ως προς τις εκθέσεις αυτές στο Συμβούλιο. και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πρόσβαση σε αυτές τις εξαμηνιές ε, εκθέσεις θα μπορούσαμε να, τις, ε, ε, να, γνωρίζουμε το περιεχόμενο και να τις εγκρίνουμε ενδεχομένως. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε το περιεχόμενο, να μας γνωστοποιείτε το περιεχόμενο των εξαμηνιαίων εκθέσεων. Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή, αλλά αυτό που θα πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι θα ήθελα μία έκθεση συνένεσης και να διαπραγματευτούμε ό,τι είναι διαπραγματεύσιο. Γνωρίζοντας τώρα ότι είμαστε ισότιμοι με το Συμβούλιο. Ελπίζω να έχουμε και μία άλλη, μία πέμπτη περίσταση να συζητήσουμε το θέμα γνωρίζοντας και τη νέα νομική βάση της Κομισιόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω ότι καταρχήν δεν αντιτίθεμαι σε αυτή την πλαισίωση. Πρόεδρος. Υπάρχει συνενετικό πνεύμα ή πνεύμα συνεργασίας για μια ενδεχόμενη συνένεση. Δεν μου ελέγχθη κατά πόσο, δεν γνωρίζω κατά πόσο η Επιτροπή θα ήθελε να παρέμβει, δεν νομίζω. Άρα τελειώσαμε με την ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί. Πολύ καλά τα νέα και θα τα πούμε στις 3 το απόγευμα. Γεια σας.